Good morning. Uh, Με, λέγομαι Άννα Γκόμες και είμαι η πρώτη αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εξ ονόματος της Υποεπιτροπής θα ήθελα να σας απευθύνω θερμό, καλώς, θερμός καλώς ορίσατε ιδίω τους συναδέλφους μας ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων καθώς και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Επίσης εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την παρουσία τους εδώ στους εμπειρογνώμονες κύριο Χάμιλτον, Ζαμπορόφσκι και Χάντονι και είναι οι εμπειρογνώμονες που ελπίζω ότι θα μας δώσουν ε, τρόφι για σκέψη με τις ιδέες που θα υποβάλουν στην συζήτηση για τις προκλήσεις και μελλοντικέ προοπτικές για την ε, διατλαντική για διατλαντικές μάλλον ε, σχέσεις και συνεργασία που πρόκειται για συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Συνέδρισης, του ε, ΝΑΤΟ. Έχουμε ε, διερμηνία σε όλες τις ε, γλώσσες εργασίες με την εξαίρεση των δανέζικων, φιλανδικών, εστονικών και βουλγαρικών. Η ακρόαση είναι προσιτή και στους πολίτες, είναι προσβάσιμη και στους πολίτες μέσω του διαδικτύου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, εξ ονόματος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το μήνυμα ότι ο Τζον Τάνερ, βουλευτής των ΗΠΑ, μας έφερε μήνυμα στην Βαλένσια πέρυσι μήνυμα του τότε υποψήφιου Πρόεδρου Ομπάμα, ο οποίος επενεί το έργο της συνέλευσης και εκφράζει την επιθυμία και πρόθεσή του να συνεργαστεί στενότερα με τις χώρες της συμμαχίας. Εμείς επιθυμούμε να υπάρχει ε, μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εποπτεία στις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και για τον σκοπό αυτό η κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ θα πρέπει να παίξει ε, σημαντικότερο και ενεργότερο ρόλο παρακολούθησης και εποπτείας των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο ΝΑΤΟ ως βήμα για, τον διατατικό διάλογο και ως εγγυητή της ασφάλειας και σταθερότητας στην Ευρώπη. Έχουμε την πρώτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, την, ε, για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ την έκθεση του Άρη Βατάνεν, την οποία εγκρίναμε προ λίγων ημερών στα μέσα Φεβρουαρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έχουν συμπήξει μια στρατηγική συμμαχία ή εταιρική σχέση αν θέλετε που έχει πια ρίξει γερές ρίζες και χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που προσφέρει το ΝΑΤΟ έχει, δίνεται πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και επίσης στην χρήση ε, νατοικών δυνατοτήτων. Και νομίζουμε ότι αυτές ε, οι πτυχές πρέπει να βελτιωθούν ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική συνεργασία μας. Πιστεύουμε επίσης ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινηθούν προς μια στενότερη συνεργασιακή σχέση λαμβάνοντας υπόψη και την διαρκή εξέλιξη της ε, πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρόσφατα ψηφίσματά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνει να αναπτυχθεί η υφιστάμενη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ με σεβασμό βέβαια της ανεξαρτησίας των δύο αυτών οργανισμών. Αυτά άλλωστε αναφέρει ως κύρια σημεία και έκθεση Βατάνεν που σας είπα πριν. Πιστεύουμε ιδίως ότι μια γνήσια συνεργασία θα πρέπει να αναπτυχθεί στο Κόσοβο και στο Αφγανιστάν. Εν προκειμένου Ζητούμε η τεχνική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, οι σχετικές συμφωνίες δηλαδή, να υπογραφούν το, δυνατότερο, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία των αποστολών μας στο Κόσοβο και στο Αφγανιστάν και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού που βρίσκεται στις αποστολές αυτές στα σημεία αυτά του κόσμου. Υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις το 2008 και θα υπάρξουν και άλλες το 2009 που πιστεύω ότι θα έχουν και σημαντικές επιπτώσεις στην σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, των δύο ε, ακτών του Ατλαντικού. Με συνεργασία με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση του ε, Πρόεδρου Ομπάμα, την, τα 60 γενέθλια του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, την εκρήου συμμετοχή της Γαλλίας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, το βάθεμα των ε, σχέσεων ασφάλειας μεταξύ Ένωσης και ΝΑΤΟ, την κύρωση της ε, ε, συνθήκης της αγώνας, την, την έναρξη συζητήσεων σχετικά με τις πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και εν τέλει, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, την μελλοντική προοπτική της αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη, το ρόλο του ουρανίου ε, και την αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη. Όλες αυτές οι εξελίξεις αναμένουμε ότι θα γίνουν μέσα στα πλαίσια μιας βαριάς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία θα αυξήσει την πίεση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και επί των ούτως ή άλλως περιορισμένων πόρων των προϋπολογισμών μας και ενδέχεται να οδηγήσουν και σε προστατευτικά μέτρα και ιδίως στις αγορές εξοπλισμών. Πρόσφατα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λάβαμε θαραλές αποφάσεις στον τομέα αυτό. Μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών εγκρίναμε οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες εξοπλισμών, η, η οποία οδηγία θα ανοίξει τις ευρωπαϊκές αγορές εξοπλισμών και ελπίζω ότι θα επιτρέψουν και στους φίλους και συμμάχους μας στο Αμερικανικό Κογκρέσο και ε, Γερουσία ότι θα σταματήσουν, θα ανακόψουν την πορεία του νόμου Buy American αποφεύγοντας έτσι τέτοια σφάλματα και θα επιτρέψουν να προχωρήσει η σύμβαση για την αγορά αεροσκαφών ανεφοδιασμού από την US Air Force. Έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και εμεί ω η μεγαλύτερη εξαγωγή εξαγωγής εξοπλισμών στην, στον κόσμο. Εμείς κάναμε ήδη νομικά δεσμευτικό τον κώδικα διοντολογία μα για τι εξαγωγέ εξοπλισμών και μαζί με τι ΗΠΑ θέλουμε να παίξουμε πρωτοπόρο ρόλο στον κόσμο στην αναζήτηση στην ε, ε, επίτευξη μάλλον της υπογραφής μιας διεθνούς συνθήκης για τον περιορισμό και την ε, νόμιμοποίηση των εξοπλισμών. Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και καλύτερο καταμερισμό των βαρών μεταξύ των μερών της συμμαχίας. Πιστεύουμε ότι η ασφάλεια και η άμυνα θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο μέσα στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη. Και γι' αυτό εκφράζουμε και την ικανοποίησή μας για το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Αμερικανών ε, για, την ευρωπαϊκή ασφάλεια με τη συμμετοχή τους σε μεγαλύτερο βαθμό στην EULEX, στο Κόσοβο, καθώς και στο Ευρωκόρ. Με τον τρόπο αυτό ανοίγουμε δρόμους για μια γνήσια σχέση μεταξύ Ενωμένης Ευρώπης και Ενωμένων χωρίς να υπονομεύουμε βέβαια το ΝΑΤΟ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο και συμπατριώτη μου αλλά και σύντροφό μου από το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ζούλιο Μιράντα Κάλια που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Άννα Μαρία, σε ευχαριστώ. Νομίζω μπορούμε να μιλήσουμε με πορτογαλικά, έτσι δεν είναι. Ε, σε ευχαριστώ για την υποδοχή σα, αγαπητοί συνάδελφοι. Στα αγγλικά και εγώ θα ήθελα να σα καλωσορίσω όλου εδώ ε, εκ μέρου ε, τη κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Επίση πρέπει να ευχαριστήσουμε το Κοινοβούλιο διότι διοργάνωσε αυτή την τόσο μεγάλη σημερινή μα συνάντηση γιατί τόσα χρόνια είναι πάρα πολύ αργαστή η συνεργασία μα με το Κοινοβούλιο και αυτό ιδίως γίνεται με ενεργή συμμετοχή της αντιπροσωπείας με, τη, με το ΝΑΤΟ. Η συνάδελφος εδώ δεξιών πάντοτε συμμετέχει και συνεργαζόμαστε με την Υποπιτροπή βεβαίως για την ε, άμυνα. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ε, περαιτέρω συνεργασία η οποία θα μας ε, βοηθήσει και θα γίνει ένα πρότυπο για τις ε, σχέσεις γενικότερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σήμερα εδώ ως ε, ε, καλεσμένοι και περιμένω πώς και πώς να ακούσω τις εισηγήσεις τους. Επίσης, θα πρέπει να σας πω για την κοινωνική μας συνέλευση ότι έχουμε 33 συλλογικά καφέ. Ε, οκτώ χώρες μέλη εκπροσωπούνται σήμερα εδώ, από την κοινωνική συνέλευση. Και σήμερα. Τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι το μέλλον των ε, υπερατλαντικών σχέσεων ε, σε επίπεδο ασφάλειας. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο, πάρα πολύ καυτό για μια σειρά λόγων. Πρώτον, έχουμε νέα κυβέρνηση στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, υπό την ηγεσία του Πρόεδρου Ομπάμα. Ήδη επομένως τα πράγματα άλλαξαν όσον αφορά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ε, αυτά τα είπε ο Αντιπρόεδρος η ε, στην ε, διάσκεψη του μονάχου τον μήνα που πέρασε. Εμείς πρόκειται να συνοηθούμε, πρόκειται να αφογκραστούμε, πρόκειται να διαβουλευτούμε με τους Αμερικανούς διότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξο τα, τα, σχέδια τα οποία έταξε αυτή η νέα κυβέρνηση και επίσης ε, είπαν ότι παραμένουν ε, ε, προσανατολισμένοι εις μια εξέλιξη των υπερατλαντικών σχέσεων. Θα πρέπει επομένω να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Μπάιντεν και σε επίπεδο ανανέωσης του ΝΑΤΟ, των σχέσεων με τον ΝΑΤΟ και πρόκειται στο Στρασβούργο να γίνει μια συνάντηση ούτως ώστε να εορταστεί η έκτη επέτειος και κατά τον τρόπο πρόκειται να κάνουμε για, αυτή την, ε, για αυτά τα 60 χρόνια τα οποία έχουν περάσει από την είδηση του ΝΑΤΟ να κάνουμε μια ε, ανασκόπηση του τι έχουμε πετύχει αλλά θα προβούμε και σε αναθεώρηση των στρατηγικών μας ε, ε, προοπτικών οραμάτων. Θα πρέπει διάφορα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Τι γίνεται με το άρθρο 5, ποια, ποια είναι η, η έννοια του σήμερα, τι προστεθεμένη αξία μπορεί να υπάρχει από τον ΝΑΤΟ όσον αφορά τις νέες προκλήσεις για την ενέργεια, την ενεργειακή ασφάλεια, για, το, ε, για τον κυβερνοπόλεμο, για την πειρατεία, τι μέλλον έχει η διεύρυνση σε επίπεδο ΝΑΤΟ, ποια θα είναι η, η βάση της εξέλιξης των μελλοντικών μας σχέσεων με την Ρωσία. Αυτές είναι μόλις ε, ορισμένες από τις ιδέες που θα πρέπει να συζητηθούν. Ταυτόχρονα, τώρα που ξεκινούμε αυτή τη διαδικασία της ανανέωσης, έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και αυτή ε, διερευνά τους τρόπους ε, για να αναβαθμίσει την ε, η πολιτική της ασφάλειας. Το 2009 θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική καμπή για την ευρωπαϊκή άμυνα και έτσι θα έχουμε διάφορες ε, κινήσεις και επιχειρήσεις. Θα ξεκινήσουμε από το Κόσοβο, θα καταλήξουμε στην Σομαλία, οπότε επίσης θα περιμένουμε και την θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη ε, Λισαβόνα. Καθώ η ΚΕΠΑ εξελίσσεται, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε επικαλύψει με τον ΝΑΤΟ, αλλά έχουμε συμπληρωματικότητα αλλά και ενίσχυση του ρόλου μας σε επίπεδο ασφάλειας. Έχουμε επομένως διάφορες προκλήσεις ε, και όλο ένα πιο σημαντικές και περισσότερες. Μέσα σε αυτή την συγκυρία επιβάλλεται να έχουμε μια ισχυρή εταιρική σχέση με την πλευρά του Ατλαντικού και για αυτό η σημερινή συζήτηση για το μέλλον του ΝΑΤΟ και την, ε, το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς ως βουλευτές θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα ε, αυτή την ε, προβληματική που έχει ε, αναπτυχθεί. Να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, και το μοναδικό αυτή η συμμαχία και είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες ασφάλειας και επομένω έτσι να εμπλακεί στην υπόθεσή μας η κοινή γνώμη. Σήμερα η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ήδη έχει ξεκινήσει αυτή τη διαβούλευση όσον αφορά το μέλλον της στρατηγικής μας ε, ε, ιδεολογικής βάσης και η συζήτηση ξεκίνησε και θα συνεχιστεί για όλα αυτά τα που σας προανέφερα οπότε έτσι θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε τελικά να εγκρίνουμε κάποιες συστάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τον ε, διάλογο, τις επαφές σε κυβερνητικό επίπεδο. Επίσης ελπίζω ότι η σημερινή μας συζήτηση. Θα βοηθήσει και ε, περιμένω πώς και πώς να ε, ακούσω την ε, σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Και σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία αυτή και σας τονίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Και αυτό θα ωφελήσει την υπόθεση ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ τώρα πάμε τώρα στο πρώτο πανελ. Οι απόψεις των ΗΠΑ όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες όσον αφορά τις διατλαντικές σχέσεις. Νταν Χάμιλτον, δόκτορα. Είστε ε, μέλος του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς. Συνεργάζεστε και με το περιοδικό ε, Foreign Policy και με διάφορα think tank. Επίσης είστε εκτελεστικός διευθυντής του Κονσόρτιουμ για τις ε, αμυντικές μελέτες στην Ουάσιγκτον. Ε, Επίσης συνεργάζεται και με το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχετε κάνει και αναπληρωτή γενικός γραμματέας της Υπηρεσίας για τη σχέση με την Ευρώπη και για τα διατλαντικά θέματα για την ασφάλεια. Επίσης έχετε ασχοληθεί και με την σταθεροποίηση στην Ανατολική Ευρώπη. Ε, διευθυντής διαμόρφωση πολιτικής, ευρωπαϊκές υποθέσεις και επίσης ε, σύμβουλος στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Γερμανία. Γράψατε πρόσφατα μία μελέτη όσον αφορά την αναγέννηση της ε, συμμαχίας του ΝΑΤΟ και συνεργαστήκατε με αυτά τα τέσσερα think tanks ούτως ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η διατλαντική, υπερατλαντική συμμαχία. Έχετε 10 λεπτά για την εισήγησή σας ε, δόκτωρα και μετά ε, έχουμε συζήτηση 15 λεπτών και όποιος θέλει όταν τελειώσει ο, ο δόκτωρ Χάμιλτον μπορεί να σίγουρα στο χέρι να στήσει το λόγο και ε, θα συντάξουμε έτσι μια λίστα αγορητών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ και βλέπω και αρκετούς φίλους. Όπως είπε η πρόεδρό θα αναφερθώ σε μία έκθεση την οποία συντάξαμε μαζί με άλλα τρία think tanks. Νομίζω ότι έχετε κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε executive summary αλλά ε, υπάρχουν έτσι και αλλιώ τα κείμενα αυτά στις ιστοσελίδες των think tank τα οποία εκπροσωπώ. Λοιπόν, τα think tank αυτά μετά από έξι μήνες διαβουλεύσεων και μελέτης και από τη μία πλευρά του Ατλαντικού και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού καταλήξαμε σε κάποιες προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές αντιλήψεις. Κάναμε συναντήσεις σε πάρα πολλές πρεσβείες ευρωπαϊκών χωρών στη Ουάσιγκτον. Συναντηθήκαμε και με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς στην ουσία αυτό το οποίο ζητάμε είναι να υπάρξει μια αναζωογόνηση της διατλαντικής στέχης ε, μένουμε λίγο στο ΝΑΤΟ επειδή θα έχουμε σύντομα τη συνάντηση κορυφής. Ζητάμε λοιπόν να αναζωογονηθεί και το ίδιο το ΝΑΤΟ. Η, ο συμπρόεδρος μάλλον είπε ότι από τη Ουάσιγκτον τις τελευταίες μέρες φαίνεται ένα νέο ύφος. Δεν είναι μόνο νέο το ύφος ε, κύριε, είναι νέες οι εποχές, είναι να το πω καλύτερα νέα η εποχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια στιγμή, μια συγκυρία η οποία είναι δεκτική μεν για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τη σχέση μας με διαφορετικό τρόπο, για να μπορέσουμε να ανατοποθετήσουμε την Δύση στα πλαίσια ε, μιας νέας ουσιαστικά διεθνούς τάξης, και έχουμε να κάνουμε με πρακτικές οι οποίες άλλοτε είναι ορθόδοξες, άλλοτε δεν είναι ορθόδοξες, είναι καινοτόμε και απαιτούν από πλευράς μας διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Λοιπόν, τι διαφοροποιεί την σχέση ε, την οποία έχουμε σήμερα από το παρελθόν και από αντίστοιχες άλλες σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές δυνάμεις. Γιατί η διατλαντική αυτή αν θέλετε σχέση συμμαχική είναι σημαντική σήμερα, παραμένει σημαντική, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό και αν ναι γιατί. Εγώ πιστεύω και εμείς πιστεύουμε ότι κατά δύο τρόπους αυτή η σχέση είναι σημαντική και δεν χαρακτηρίζει με τον ίδιο τρόπο καμιά άλλη διεθνή σχέση ανάμεσα σε δύο μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις. Καταρχάς, τις τελευταίες έξι δεκαετίες έχουμε σωρεύσει υλικό, έχουμε σωρεύσει κεφάλαιο στα πλαίσια των σχέσεών μας. Αυτό φαίνεται και σε σχέση με αυτό που ονομάζετε εσείς το ακή κομινοτέρ, το κοινοτικό και εκτιμένο. Είναι κάτι το οποίο είναι το ομόλογο αν θέλετε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε ένα αντίστοιχο τέτοιο ακί, ένα αντίστοιχο τέτοιο κεκτημένο το οποίο θα το ονόμαζα όχι ακί κομινοτέρα αλλά ακί ατλαντικ. Έχουμε συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας, συγκεκριμένες μορφές διαβούλευσης που έχει δημιουργήσει τελικά κάτι το οποίο μπορεί να είναι λίγο άμορφο αλλά είναι κάτι που διαφοροποιεί τις σχέσεις μας από σχέσεις άλλων δυνάμεων στον κόσμο φροντίζουμε οι μεν τους δε, φροντίζουμε ο ένας τον άλλο. Για πολλές δεκαετίες πάντα εμείς τιμήσαμε το λόγο μας αν θέλετε, τη σχέση τη φιλική την οποία πάντα είχαμε. Έχουμε μια ελεύθερη σχέση και αυτή τη σχέση πρέπει να συνεχίσουμε να την καλλιεργούμε. Έχουμε προσδοκίες οι οποίες δεν είναι φυσικά στο ίδιο επίπεδο των επιτευγμάτων μας. Παρόλα αυτά οι προσδοκίες μας είναι τέτοιες που μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε εφόσον εμείς βέβαια το επιθυμούμε να το κάνουμε. Δεύτερον, στον κόσμο σήμερα, αν μια διεθνή συμμαχία θέλει να είναι αποτελεσματική, πρέπει να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είμαστε, αν θέλετε, ο πυρήνας ή ασδήποτε μορφής διεθνούς συμμαχίας Είμαστε απαραίτητοι. Είμαστε βέβαια απαραίτητοι αλλά δεν είμαστε επαρκείς από μόνοι μας. Αν τυχόν υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, στην ουσία καθιστούμε η αδίποτε σφαιρική παγκόσμια συμμαχία αναποτελεσματική δεν έχουμε άλλου είδους τέτοιες ε, σχέσεις ε, με άλλους εταίρους. Όπως είπε ο Τζο Μπάιντεν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υλικό, το οικοδομικό που έχουμε και να χτίσουμε αυτή τη σχέση που έχουμε. Αν θέλουμε όμως μπορούμε να μην το κάνουμε και μπορούμε να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε σαν παιδιά για το βοδινό κρέας, για τις ορμόνες, για τις μπανάνες και για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Προφανώς και έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις Έχουμε το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Αλλά ο παγκόσμιος πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας έχει τελειώσει εγώ νομίζω. Έχουμε προβλήματα διμερών συγκρούσεων. Αυτό δεν έχει απομακρυνθεί. Αλλά παρόλα αυτά οι μεγάλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή λειτουργούν εν ειρήνη και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Πέραν αυτών των ορθοδόξων αν θέλετε διακυβερνητικών σχέσεων έχουμε και μη ορθόδοξες πρακτικές στη διεθνή σκηνή που μας δημιουργούν προκλήσεις. Νομίζω ότι δεν είμαστε απόλυτα εξοπλισμένοι να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε κάποιες στρατηγικές προκλήσεις οι οποίες αμφισβητούν τη σχέση μας και η πρώτη πρόκληση είναι αυτό που ονομάζουμε γενικά οικονομική κρίση. Τα χρηματοπιστωτικά όπως επίσης ε, και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε άλλους τομείς όπως η ενέργεια είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Η συμφωνία την ομάδα των 20 είναι κάτι που θα περιλαμβάνει και τις συμφωνίες στις οποίες εμείς καταλήγουμε ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Έχουμε και άλλες στρατηγικές προκλήσεις οι οποίες επαναλαμβάνω δεν είναι ιδιαίτερα ορθόδοξες. Να πω ένα πράγμα μόνο ε, κάτι το οποίο θεωρήθηκε μη ορθόδοξο, αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς αντοχή. Από κοινού οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν μία σειρά προκλήσεων οι οποίες δεν είναι εύκολα θα έλεγα περιγράψιμες και περιλήψιμες στα πλαίσια μίας παραδοσιακής πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας. Σαν παράδειγμα, έγκλημα στον κυβερνοχώρο από τη μία, αλ από την άλλη. Υπάρχουν δίκτυα και από τη μία, υπάρχουν δίκτυα και από την άλλη τα οποία υπονομεύουν τις ελεύθερες κοινωνίες. Ε, προσπαθούν όχι να κατακτήσουν εδάφη με την έννοια την παραδοσιακή του πολέμου, αλλά χρησιμοποιούν τα μέσα της ελεύθερης κοινωνίας, τα διαθέσιμα μέσα για να αμφισβητούν τη συγκεκριμένη κοινωνία. Αυτό δημιουργεί σε πάρα πολλές ανομαλίες και μερικές φορές και σε καταστροφές. Και δεν είμαστε εξοπλισμένοι με τον κατάλληλο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές, είτε σε διεθνές επίπεδο, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε σε επίπεδο μεγαλύτερη Έχουμε πολλά προβλήματα με τα οποία ασχολούμαστε όπως το θέμα των ονομάτων των επιβατών κτλ. Το πρόβλημα είναι όμως πώς θα προστατεύσουμε τις κοινωνίες μας απέναντι σε αυτές τις νέες απειλές και πώς θα καταστήσουμε τις κοινωνίες μας ανθεκτικές και μη επηρεάσιμες από τις νέες αυτές απειλές. Ο βασικός χώρος για να το κάνουμε αυτό είναι οι διμερείς επαφές, οι διεθνείς επαφές, και φυσικά και οι επαφές ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εντοπίσει πάρα πολλούς τομείς στους οποίους θα μπορέσουμε να παίξουμε πολύ συγκεκριμένο ρόλο και μέσω του ΝΑΤΟ. Πολύ συγκεκριμένο ρόλο, περιορισμένο ίσως αλλά σημαντικό. Αν δείτε λοιπόν τα έγγραφα τα οποία έχουμε ετοιμάσει, πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα είναι επαρκή σαν μέσα. Η απάντηση είναι απλή, όχι πρέπει να αναρρυθμίσουμε για μια ακόμη φορά τους νέους μηχανισμούς για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του νέου κόσμου. Και η σχέση ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ένωση είναι σημαντική. Έχουμε άμεσα προβλήματα, Αφγανιστάν από τη μία, Ρωσία από την άλλη, διαφορετικά προβλήματα διαφορετικού επίπεδου βέβαια, αλλά απαιτούν και τα δύο, καλούν και τα δύο συνοχή ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και κοινή δράση θα επανέλθουμε στις λεπτομέρειες, αλλά αυτά τα δύο προβλήματα δεν περιμένουν, είναι άμεσα προβλήματα. Αν κοιτάξετε επίσης ε, γενικότερα τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα και εγώ ήμουν από αυτούς που είχε προωθήσει την ιδέα από το 1995 το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα σήμερα, κινείται η σχέση αυτή σήμερα, θα το χαρακτήριζα δυσλειτουργικό και ανεπαρκές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή όμως η δυναμική να δημιουργήσουμε ένα βελτιωμένο πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο να είναι πιο στρατηγική. Στρατηγικό το πλαίσιο γιατί οι σχέσεις μας δεν είναι επαρκώς στρατηγικές και αν θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα μέσω του ΝΑΤΟ, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχύσουμε τη σχέση μας. Ζητάμε λοιπόν να υπάρξει μια νέα διαδικασία στον τρόπο αντιμετώπισης και χάραξης του πλαισίου των σχέσεών μας, ο οποίος να ξεπερνά την εμβέλεια των σημερινών. Για το ΝΑΤΟ πιο συγκεκριμένα. Αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι το εξή. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ΝΑΤΟ είναι ο τερματισμός του ψυχρού πολέμου και δεν πολέμησε ποτέ το ΝΑΤΟ σαν τέτοιο, έτσι δεν είναι για όλες αυτές τις δεκαετίες. Σήμερα το ΝΑΤΟ εμπλέκεται σε πέντε αποστολές. Είναι πιο απασχολημένο από, πετέ, από ποτέ. Παρόλα αυτά όμως ο κόσμος δεν δίνει σημασία στο ΝΑΤΟ. Οι κυβερνήσεις δεν δίνουν σημασία στο ΝΑΤΟ. Λόγω διαφορετικών αντιλήψεων, διαφορετικών πολιτικών πολιτισμών, διαφορετικών παραδόσεων Παρ' όλα αυτά εμπλέκεται το ΝΑΤΟ σε πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα στον τομέα της διεθνούς ασφάλειας, αλλά δεν πετυχαίνει να τα λύσει προς το παρόν. Είναι πιο απασχολημένο και πιο δραστήριο από ποτέ το ΝΑΤΟ σήμερα. Παρ' όλα αυτά δεν απασχολεί ούτε τα κοινοβούλια, ούτε τις κυβερνήσεις για το ποια θα είναι η νέα λογική και το νέο σκεπτικό λειτουργίας του. Απαιτείται λοιπόν εμείς να αντιμετωπίσουμε με στρατηγικό τρόπο τη σχέση μας με το ΝΑΤΟ. Σε δύο φάσεις το προβλέψουμε αυτά να δημιουργήσουμε καταρχάς μια επιτροπή σε επίπεδο κλιμακίων του ΝΑΤΟ και να υπάρξουν ε, κάποιες προτάσεις για τη νέα αρχιτεκτονική και για το πώς θα ταιριάζει το ΝΑΤΟ στις κοινέ παγκόσμιες προσπάθειες στο μέλλον. Και δεύτερο να περάσουμε και σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις του ΝΑΤΟ αυτή η task force θα κάνει προτάσεις στους υπουργούς και στις κυβερνήσεις και στο στρατηγείο στις Βρυξέλλες έτσι ώστε να γίνουν κάποιες τελικές προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές από το Υπουργικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ ή από τη συνάντηση κορυφής ή έστω το 2010. Αυτές είναι οι προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Αν δείτε το τι είναι το ΝΑΤΟ σήμερα. Απαιτεί μια νέα εσωτερική ισορροπία. Για 15 χρόνια είπαμε ότι ή θα πάμε και εκτός χώρου ή θα κλείσουμε το μαγαζί. Παρ' όλα αυτά εμείς είμαστε εκτός χώρου. Φύγαμε από την Ευρώπη και το βορειοατλαντικό χώρο. Είμαστε στο Χιντουκούς. Αλλά μόνο ε, δεν το κλείσαμε το μαγαζί. Σε καμία περίπτωση δεν έγινε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει η δύναμη την οποία χαρακτηρίζουμε πάρα πολύ απλά σαν τη δύναμη που μας προστατεύει και μπορούμε να πείσουμε εύκολα τον κόσμο, όχι πολύ εύκολα βέβαια, ότι το να είμαστε στο Χίντου Κούσου σήμερα είναι ένα κομμάτι αυτής της προσπάθειας προστασίας της Ευρώπης και την ΝΥΠΑ σήμερα. Το ΝΑΤΟ όμως δεν είναι και τόσο ορατό βέβαια στα πλαίσια των νέων του στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Είναι ορατό το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, δεν είναι ορατό στην Ευρώπη. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Αυτή η διαφορά είναι σημαντική διαφορά και δημιουργεί προβλήματα. Αν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τον δικό μας χώρο, πώς θα προβλέψουμε και πώς θα αναπτύξουμε τις δυνάμεις μας αλλού. Ζητάμε λοιπόν μια νέα υπηρεσία ανάμεσα στις εσωτερικές δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και στις εξωτερικές δραστηριότητες. Εσωτερικές απλές τρία πράγματα. Πρώτον συλλογική άμυνα, η προηγούμενη αποστολή της Υπάρχουν νέα μέλη στο ΝΑΤΟ και αναρωτιόνται ε, για την αξιοπιστία θα έλεγα των εγγυήσεων του άρθρου 5. Άλλες χώρες θεωρούν ότι όλα αυτά είναι υπερβολές. Αλλά λέγεται ότι αν έστω και μία χώρα πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά μια απειλή, γιατί αυτό σημαίνει αλληλεγγύη, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις εγγυήσεις που έχουμε γύρω από την εφαρμογή και τη λειτουργία του άρθρου 5 και θα πρέπει να υπάρξουν ε, νέες προτάσεις και προγραμματισμοί για την χρήση του άρθρου 5, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα γίνονται συνεχώς ασκήσεις σαν παράδειγμα στρατευμάτων υπό την καθοδήγηση του ΝΑΤΟ, υπό την ε, διοίκηση του ΝΑΤΟ, αλλά δεν ονοματίζονται ποτέ σαν ασκήσεις του ΝΑΤΟ, ονοματίζονται σαν διμερείς ασκήσεις ή πολυεθνικές ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Υπάρχουν και, και άλλοι τομείς στους οποίους το ΝΑΤΟ μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Σαν παράδειγμα οι περιοχές της βορειοατλαντικής περιοχής οι οποίες χρήζουν ελέγχου. Στο Μεσόγειο υπάρχει η δυνατότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 5. Εμείς εμποδίζουμε δηλαδή μέσω ναυτικών επιχειρήσεων κάποια απαράδεκτα προϊόντα να φτάνουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν ρόλοι για το ΝΑΤΟ στον τομέα της ενίσχυσης της αντοχής της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και στον τομέα του βιολογικού πολέμου και στον τομέα του πολέμου στον κυβερνοχώρο και ο τρίτος τομέας στον οποίο είναι σαφής η αποστολή ε, του ΝΑΤΟ είναι μια ειρηνική Ευρώπη. Αυτός ήταν πάντα ένας ιστορικός μας στόχος και δεν τον έχουμε απόλυτα πετύχει. Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, η Ευρώπη που έχουμε σήμερα δεν είναι η Ευρώπη την οποία θα θέλαμε. Ο χώρος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ρωσία είναι ένας χώρος φεός ουσιαστικά. Κι όμως εκεί το μέλλον είναι ιδιαίτερα προβληματικό και πρέπει να τους βοηθήσουμε τους κατοίκους των περιοχών αυτών για να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Είχαμε προβλήματα μετά από μεγάλες τραγωδίες στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για χώρους οι οποίοι ήταν στρατηγικοί και για τις Ηνωμένε Πολιτείες και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω ότι σαν ΝΑΤΟ θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασικές αποστολές, ξεκάθαρες αποστολές, προσπαθούμε να ανταεξηγήσουμε αυτά που πρέπει να κάνει το ΝΑΤΟ στο κοινό και έχουμε και τις αποστολές εκτός Ευρώπης με την δυνατότητα ανταπόκρισης μέσω των δυνάμεων επέμβασης που έχει στη διάθεσή του το ΝΑΤΟ. Μπορούμε να προβάλλουμε την δυνατότητα επιχειρήσεων σε μεγάλη απόσταση όπως το Αφγανιστάν. Ποιος ξέρει πώς θα εξελιχθεί η δυνατότητα αυτή. Είδαμε ότι και στα Βαλκάνια και στο Αφγανιστάν ότι όταν κάνει κάτι το ΝΑΤΟ υπάρχουν συνήθως ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται για δυνάμεις σταθεροποίησης. Το ΝΑΤΟ εδώ δεν ηγείται των προσπαθειών σταθεροποίησης. Παρ' όλα αυτά πρέπει να έχει συγκεκριμένες δεδομένες επιχειρησιακές δυνατότητες για να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Και μια τελευταία αποστολή εκτός Ευρώπης. Αν μοιράσουμε τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ σε πάρα πολλές αποστολές πρέπει να προσέξουμε για να μην το διαρρήξουμε σε εισαγωγικά το ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να το τεντώνουμε τόσο πολύ. Πρέπει να είναι το ΝΑΤΟ ικανό να δουλεύει καλά σε σωστή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες που παρέχουν δυνάμεις να παρέχει τις σταθεροποιητικές δυνατότητες και τις δυνατότητες εγγύησης ασφάλειας τις οποίες πρέπει να παρέχει. Αυτό που κάνουμε στην έκθεσή μας εμείς λοιπόν είναι να υπογραμμίζουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί στα πλαίσια μιας στρατηγικής σχέσης αν ξεπεράσουμε κάποια μικρά εμπόδια, κάποια εμπόδια μάλλον. Με φάνταστο τρόπο προσπαθούμε να προβάλλουμε το τι μπορούμε μαζί να κάνουμε όπως κοινέ προμήθειες, κρίση, ε, διαχείριση κρίσεων εφόσον ξεπεράσουμε κάποια άλλα προβλήματα τα οποία μας μπλοκάρουν το ΝΑΤΟ και, το, και τα Ηνωμένα Έθνη υπέγραψαν μια συμφωνία την προηγούμενη, ε, την προηγούμενο φθινόπορο. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή σε επίπεδο κοινή γνώμη αυτό δεν έπρεπε να γίνει ιδιαίτερα δεκτό, γιατί δημιουργούνται προβλήματα. Και εν πάση περιπτώσει το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη σε χώρες όπως το Αφγανιστάν σαν παράδειγμα πρέπει να είναι εταίροι σημαντικού επίπεδου. Υπάρχουν και άλλοι θεσμοί βέβαια με τους οποίους πρέπει να αναπτυχθούν οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ. Αυτά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δούμε για τον ΝΑΤΟ και τρεις βασικές αποστολές ε, στο εσωτερικό του χώρου του ΝΑΤΟ και τρεις βασικές αποστολές στο εξωτερικό του χώρου. Ακόμα και οι εσωτερικές αποστολές απαιτούν δυνάμεις επιχειρησιακές. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να επανεξετάσει τις δυνατότητες που έχει και να ακυρώσει ό,τι το στάσιμο και στατικό περιλαμβάνει. Θα κάνουμε προτάσεις και για τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, τις έχετε σε λεπτομέρειες ε, στον φάκελό σας. Πρώτον, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον κανόνα της συνένεσης στο ΝΑΤΟ, όχι να τον καταργήσουμε. Ε, θα πρέπει να υπάρχει συνένεση για τις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και για τα οικονομικά. Όταν όμως πάρουμε κάποια απόφαση και κάποιες χώρες μόνο πάρουν μέρος στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αυτές θα πρέπει να αποφασίζουν για το πώς θα εξελιχθεί η επιχείρηση. Οι χώρες οι οποίες έχουν συμφωνήσει με την επιχείρηση αλλά δεν συμμετέχουν σε αυτή δεν θα πρέπει να παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο. Κάνουμε προτάσεις και για τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου το North Atlantic Council μερικές φορές μπλοκάρεται από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Γιατί να μην υπάρξει λοιπόν ένας τροποποιημένος τρόπος εφαρμογής της αρχής της συνένεσης τουλάχιστον στις χαμηλότερες, στα χαμηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν δύο στρατηγία στο ΝΑΤΟ, ένα στη Βόρεια Βιρτζίνια και ένα εδώ στο Βέλγιο, με δύο στρατηγούς. Εμεί πιστεύουμε ότι το ACT του Norfolk στη Βόρεια Βιρτζίνια θα πρέπει να έχει σαν διοικητή Ευρωπαίο. Θα πρέπει να ανασχεδιαστεί, να υπάρξει μια νέα ισορροπία και να υπάρχει ε, δυνατότητα ευρωπαϊκής παρέμβασης και μέσω της κοινή διοίκησης ή της συνδιοίκησης από το στρατηγείο του Norfolk. Έτσι θα αναπτύξουμε περαιτέρω δυνατότητες από αυτές που έχουμε σήμερα διαθέσιμες. Θέλουμε επίσης και τρία κοινά στρατηγία στις Βρυξέλλες, στην Ολλανδία και μία στη Λισαβόνα. Κάθε ένα από τα στρατηγία αυτά θα έχει έναν τομέα γεωγραφικό στον οποίο θα ειδικεύεται και τα στρατηγία αυτά θα ελέγχουν επίσης και τις έκτακτες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα διαβάσετε παρακαλώ, να τα σχολιάσετε και πέραν της περιλήψεως την οποία σας παρέχουμε νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ειδικέ προτάσεις για την πυραυλική άμυνα, για τις πυρηνικές δυνάμεις αλλά αυτά είναι θέματα που ίσως θέλετε να τα συζητήσουμε καλύτερα για να μην μακρηγορώ. Σας ευχαριστώ. Την προηγούμενη εβδομάδα με μια μικρή αλλά εκλεκτή αντιπροσωπεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο, Κοινοβούλιο είχαμε, βρεθήκαμε στην Ουάσιγκτον για μια fact-finding mission για να δούμε τι πρόκειται να προσφέρει η νέα Αμερικανική κυβέρνηση στο μέλλον. Η συνολική εντύπωση που αποκομίσαμε ήταν πολύ ενθαρρυντική και κυρίως για θέματα όπως έλεγχος των εξοπλισμών, αφοπλισμός, ε, ισχυρή δέσμευση για σημαντική μείωση των στρατηγικών πυρηνικών όπλων, πράγματα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά για να αυξήσουν την αξιοπιστία όταν μιλούμε για θέματα όπως μη διασπορά των πυρηνικών όπλων και νομίζω ότι όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και σημαντικά. Επίσης μας άρεσε η προθυμία που διαπιστώσαμε για άμεσες ε, διαβουλεύσεις με το Ιράν για το θέμα το πυρηνικό. Δεν ανοίγει κανεί όλα τα χαρτιά του βέβαια από την αρχή στις διαπραγματεύσεις, αλλά ένα θέμα που απεκόμισε ως εντύπωση από τις συζητήσεις αυτές είναι ότι μου φαίνεται ότι κάθε φορά που οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι μιλούν για το Ιράν, οι Αμερικανοί το μόνο που καταλαβαίνουν είναι κυρώσεις. Εμείς θα θέλαμε να αρχίσουν να σκέπτονται οι Αμερικανοί και τη λέξη κίνητρα. Μια παράλληλη προσέγγιση που δεν αρκεί βέβαια να γράφεται στα χαρτιά, πρέπει να βρει εφαρμογή και στην πράξη. Το δεύτερο που μας ανησυχεί κάπως είναι ότι δεν υπάρχει σαφής προοπτική ακόμη σε ό,τι αφορά την κύρωση της Comprehensive Ban Treaty, της ε, συνολικής ε, συνθήκης για την απαγόρευση εξοπλισμών. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό για να αρχίσει η προσπάθεια για την μη διασπορά. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι θα μπορέσετε να πείσετε αρκετούς ε, γερουσιαστές, να πιστούν εν πάση περιπτώσει αρκετοί γερουσιαστές, ώστε να κυρώσουν τη συμφωνία αυτή. Δεν θα αναφερθώ τόσο πολύ σε αυτά που είπατε για το ΝΑΤΟ, γιατί αυτό ας το κάνουν καλύτερα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Εγώ σκέπτομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται περισσότερο με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν πολλά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να συζητηθούν άμεσα στις σχέσεις με τις ε, Ενωμένες Πολιτείες. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε ταχθεί υπέρ ενός άμεσου διαλόγου ασφάλειας με τις ΕΠΑ Πολιτείες στους τομείς εκείνους όπου διαθέτει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, αποκατάσταση της αξιοπιστίας σε σχέση με τις δυτικές αξίες ε, και αυτό εντάσσεται κάπως και σε αυτή την ανθεκτικότητα της κοινωνίας που αναφέρατε εσείς. Από την άλλη μεριά έχουμε πράγματι εμπειρία στην πράξη, έχουμε και μηχανισμούς για την δημιουργία ε, μη στρατιωτικών αποστολών αλλά και αποστολών ανοικοδόμησης και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιθυμεί να διδαχθεί από μας. Γιατί λοιπόν να μην ξεκινήσουμε έναν επίσημο διάλογο ασφάλειας στους τομείς αυτούς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει και ε, νομικές αρμοδιότητες. Τελευταίο σχόλιο. Μαθαίνω, και αυτή την εντύπωση απεικόμισα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ακόμη οι Αμερικανοί όταν μιλούν για υπερατλαντικές σχέσεις εστιάζουν κυρίως μέσω του ΝΑΤΟ και σε διμερείς σχέσεις με τις ε, χώρες, με, τις, συγκεκριμένα κράτη. Αυτό είναι, εν πάση περιπτώσει, μια πραγματικότητα. Μπορεί να αλλάξει όμως αυτή η πραγματικότητα. Εσείς αναφερθήκατε σε ορισμένα θέματα όπου λέτε ότι το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα και στις σχέσεις με την άλλη ακτή του Ατλαντικού. Συμφωνώ. Τι μπορεί να γίνει από τη δική μας πλευρά, ρωτώ τώρα, για να αυξήσουμε την συνειδητοποίηση από τη δική σας πλευρά, του Ατλαντικού, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημασία για συνεργασία για κοινά συμφέροντα. Μιλήσατε για παράδειγμα για την δυνατότητα να αλλάξουν οι ε, κανόνες της συνένεσης στο ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα εδώ η συνθήκη η Ευρωπαϊκή Συνθήκη μπορεί να αποτελέσει ένα υπόδειγμα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εμείς ώστε να αυξήσουμε την συνειδητοποίηση από τη δική σας την πλευρά μεταξύ της ε, πολιτικής ελίτ αλλά και των διαφόρων think tank. Ο κύριος Λαμάλφα θα μιλήσει τώρα. Οι συνάδελφοι που θα λάβουν μετά από τον κύριο Λαμάλφα τον λόγο ας περιοριστούν στα δύο λεπτά για να μην χάσουμε περισσότερο χρόνο. Νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά που μπορούμε να ακούσουμε την ε, παρουσίαση αυτής της πολύ σημαντικής νέας έκθεσης και συγχαίρω τον κύριο Χάμιλτον που τη συνέταξε. Ίσως, κυρία Πρόεδρε, να πρέπει να συζητήσουμε την έκθεση αυτή σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας αξίζει τον κόπο να εγκύψουμε περισσότερο στο κείμενο αυτό. Η ερώτηση μου έχει σχέση με τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ γεννήθηκε ως αντίδραση σε μια απειλή που προερχόταν από την Σοβιετική Ένωση τότε. Ωστόσο, ακόμη τώρα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η σχέση με τη Ρωσία τώρα. Εάν κοιτάξουμε την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ θα δούμε ότι έχουμε διαφορετικές ευαισθησίες από τους συναδέλφους μας εμείς εδώ από αυτούς που βρίσκονται εκεί. Βρίσκουν, ε, βλέπουν διαφορετικά τη Ρωσία από ότι εμείς ε, που εμείς πιστεύουμε σε μια, ε, πιο, σε μια σχέση μεγαλύτερη συνεργασία με τη Ρωσία. Λέτε εσείς απλώς ότι χρειαζόμαστε μια ε, διπλή παράλληλη στρατηγική για τη σχέση με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο κόνσεπτ, μια νέα αντίληψη για τη σχέση με τη Ρωσία, αν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει πρώτα τι περιμένουμε από αυτήν. Ο κύριος Φλούγερ. Το έγγραφο που παρουσιάσατε έχει πραγματικά μεγάλη σημασία. Εγώ το διάβασα με μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι εντάσσεται και στην ε, παράδοση των εγγράφων του κυρίου Νάουμαν και Σακασβίλη. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες αλλά υπάρχουν και ορισμένες διαφορές. Πρόκειται πάντως για κεντρική σημασία έγγραφο για την ανάπτυξη νέας στρατηγικής του ΝΑΤΟ. Όμως το έγγραφο δεν μου αρέσει, το λέω εξ αρχής και το λέω καθαρά. Κάτι που με εκπλήσει είναι η πρότασή σας για την άρση της αρχής της συνένεσης. Γράφετε στο εγγραφό σας ότι είναι σημαντικό σύμβολο του ΝΑΤΟ αυτή η αρχή της συνένεσης. Αλλά de facto η πρότασή σας καταλήγει στην ενίσχυση των μεγάλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ και στην αποδυνάμωση των μικρών. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα Ίσως κάτι τέτοιο να έχει νόημα, αλλά ωστόσο υπονομεύει τις δημοκρατικές διαδικασίες. Άλλο που με ενδιέφερε είναι η πρότασή σας για ένα opt-out. Δηλαδή, κάποιες χώρες μέλη να μην συμμετέχουν σε ορισμένες, ε, σε αποστολές, αλλά τότε να μην έχουν και δικαίωμα να εκφράζουν άποψη. Και αυτό θίγει τη δημοκρατία και θεωρώ ότι είναι προβληματικό. Οι ερωτήσεις μου που έχω να σας απευθύνω αναφέρονται σε μελλοντικέ αποστολές που αναμένετε εσείς. Αφενός, πώς θεωρείτε ότι θα συνεχιστεί η αποστολή στο Αφγανιστάν, ποιες επιλογές ενδεχομένως υπάρχουν, δηλαδή θα συνεχίσει καταστολή των εξεγέρσεων, θα ε, γίνει ακόμα πιο έντονη η στρατιωτική παρέμβαση εκεί. Κάπως έτσι φαίνεται να κινείται η Ουάσιγκτον από ό,τι μαθαίνω. Και δεύτερο, σε ποιες περιοχές του κόσμου αναμένεται να γίνουν νέες αποστολές ή ποιες μορφές αποστολών. Για παράδειγμα, εσείς προτείνετε μια σταθεροποιητική δύναμη του ΝΑΤΟ. Άρα εδώ ρωτώ ποια μορφή θα λάβουν οι αποστολές αυτές και σε ποιες περιοχές του κόσμου θα αναπτυχθούν. Στο μόνο όπου συμφωνώ μαζί σας είναι το άρθρο της ιδρυτικής, της συνθήκης του ΝΑΤΟ ότι αυτό έχει αποδυναμωθεί και αποδυναμώνεται διαρκώς. Διότι υποτίθεται ότι η ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία και αυτά που κάνει τώρα το ΝΑΤΟ δεν έχουν σχέση με άμυνα. Και εν τέλει, μια μικρή επισήμανση, όταν λέτε ότι θέλετε a ε, home missions, τουλάχιστον ε, στο γερμανικό πλαίσιο, δεν ακούγεται καθόλου καλά αυτό, διότι αυτό θυμίζει στρατιωτικέ παρεμβάσει στο εσωτερικό τη επικράτειας μια χώρα. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν μα ηχεί καθόλου καλά. Ο κ. Βαν από την Τουρκία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Χάμιλτον για τις νέες ιδέες πολύ ενδιαφέρουσες που ακούσαμε. Να κάνω δύο σχόλια, μάλλον να θέσω μια ερώτηση και ένα σχόλιο. Στην έκθεση αυτή Σωστά αναφέρεστε στο ότι οι νέες προκλήσεις, οι σημερινές προκλήσεις απαιτούν ευρύτερε μορφές συνεργασίας. Προτείνεται επίσης νέους θεσμικούς μηχανισμούς για τη λειτουργία της διατλαντικής σχέσης. Μέχρι τώρα το ΝΑΤΟ ήταν ο βασικός μηχανισμός αυτών των σχέσεων. Μπορείτε να μας πείτε σε τι θεσμούς αναφέρεστε, τι είδους θεσμούς θέλετε να προτείνετε. Δεύτερον, και αυτό το έθεσαν και οι Γερμανοί συνάδελφοι, τροποποίηση του κανόνα του συνένεσης. Νομίζω ότι η συνένεση είναι αυτή η οποία κρατάει συνεκτικά το ΝΑΤΟ. Η αλληλεγγύη, η σενοχή διασφαλίζονται μέχρι τώρα και ε, εξαρτώνται θα έλεγα από τον κανόνα της συνενέσεως. Αν τυχόν αλλάξουμε σε βάθος τον κανόνα αυτό, φοβάμαι ότι το ΝΑΤΟ που ξέραμε δεν θα υπάρχει πια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ο κύριος Σονισκίεβιτς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Εδώ και αρκετά χρόνια οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες ήσαν εντελώς διαφορετικές από αυτές τις οποίες ελπίζουμε να είναι στο μέλλον. Για τα θέματα της ασφάλειας, αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι ότι στα πλαίσια της αμερικανικής στρατηγικής δεν υπήρχε ουσιαστικά αναφορά στο ΝΑΤΟ. Και πάνω κάτω το ίδιο βέβαια συνέβαινε και από πλευρά της Ευρώπης. Το ΝΑΤΟ το αναφέραμε μόνο περιθωριακά, περιφερειακά. Από ό,τι φαίνεται, οι βασικές αρχές της σχέσης μας στον τομέα της ασφάλειας είναι το αδιέρετο της ασφάλειας και των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Κάτι το οποίο είχαμε αγνοήσει για πολλά χρόνια, αλλά κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να μπαίνει σε μια πορεία αποκατάστασης. Πώς λοιπόν θα μπορούσατε εσείς να ανταποκριθείτε στην έκκληση της Madeleine Albright σύμφωνα με το, όχι, με το decoupling, το discrimination και το duplication, τα τρία D δηλαδή. Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στην έκκληση αυτή και πώς μπορούμε έτσι να ενισχύσουμε τη δομή του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι και εσείς υποστηρίζετε ε, πράγματι ο Σασέρ στην ε, Ευρώπη θα πρέπει να είναι Αμερικανός και ταυτόχρονα να είναι ε, και ηγέτης των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Θέατρο. Τώρα βέβαια τα προβλήματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη, βρίσκονται σε τομείς οι οποίοι είναι υπό τον έλεγχο του λεγόμενου Central Command. Πώς λοιπόν θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του ΣΑΣΕΡ και πώς θα καταστήσουμε τις δυνάμεις που ελέγχει πιο αποτελεσματικές. Το δεύτερο θέμα είναι η Ρωσία. Ξέρουμε όλοι ότι ο πρόεδρος Μετβέντεφ ξαφνικά άρχισε να προωθεί ένα θα έλεγα ομιχλώδες σχέδιο για την εκ νέου καταγραφή των σχέσεων στα πλαίσια μιας νέας δομής στον τομέα της ασφάλειας. Υπάρχουν κάποιες τάσεις από πλευράς της ασφαλείας έτσι ώστε να προωθήσουν τις προτάσεις αυτές στα πλαίσια ενός διαλόγου ξεχωριστά με την Ευρώπη και ξεχωριστά με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό είναι επικίνδυνο. Νομίζω ότι θα πρέπει εμείς σαν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί να έχουμε ένα κοινό μέτωπο. Προφανώς ο διάλογος θα πρέπει να ολοκληρωθεί ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές με τη Ρωσία. Και ο Σαρκοζή είχε δίκιο όταν λέει ότι οι συζητήσεις με τη Ρωσία θα πρέπει ίσως να γίνουν στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαλοδίσκη ονομάζομαι είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι το μέλλον του πλανήτη βρίσκεται στην αποτελεσματική συνεργασία που θα είναι και μακρόπνοη μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν τώρα λέω αφετηρία τη διατύπωση του δόκτωρος Χάμιλτον, τον οποίο και ευχαριστώ για την τόλμη, την ακρίβεια των ισχυρισμών του. Είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβανόμεθα. Ότι για τον κόσμο έχουμε υποχρέωση προστασίας και παρχής ασφάλειας. Και υπάρχει εδώ κάποια δύσκολη αντίθεση. Υπάρχει ένα δύσκολο πρόβλημα να επιλύσουμε, δηλαδή το παζλ της σχέσης μας με την Ρωσία. Για να κάτσουμε να λάβουμε υπόψη τι γίνεται με αυτό το τόξο της ε, ε, Ρωσίας. Κεντρική Ασία, Κάυκασος, ε, μετά Βαλτικές χώρες, Φινλανδία, Ουκρανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έτσι διαμορφώνεται η μεθόριος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οπότε θα πρέπει τώρα να κάτσουμε να λάβουμε υπόψη πώς θα παίξουμε αυτό μας τον ρόλο προστασίας και ασφάλειας. Είναι πολλοί οι Ρώσοι οι οποίοι κατοικούν εκείθεν αυτών των συνόρων. Και έχουμε προβλήματα και στον Κάφκαζο και στις βαλτικές χώρες. Κατά την ε, κρίση και τον πόλεμο στη Γεωργία αυτό ε, κατεφάνει. Τι θα γίνει. Θα επικαλυστούμε το άρθρο 5 επειδή κάποιος επιτέθηκε σε κάποιο χωριό. Κάποιος, Ρώση ή κάποιος άλλος. Αρκεί αυτό. Αν όμως δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, εάν δεν το πάρουμε στα σοβαρά το ρόλο μας τότε κάθε περίπτωση ε, επίθεσης και επιθετικότητας τι θα γίνει ε, υπάρχει ασφάλεια υπάρχει, υπάρχει εκπλήρωση του ρόλου μας για την προστασία να τι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ούτως ώστε αυτός ο χώρος μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης να διέπεται από αυτήν την συνεργασία που είπαμε Άρα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί για να είμαστε και σωστοί στην προστασία της ασφάλειας. Σε ευχαριστούμε κύριε Βιολοβίσκη λέει η Πρόεδρος και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καλαμπουίχ από την Ισπανία. Άννα σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο καθηγητή ο οποίος ε, ήρθε εδώ με αυτή την έκθεσή του, την εισήγησή του Βεβαίω θα πρέπει και να χαιρετήσουμε την αλλαγή αυτή που έλαβε χώρα στι ΗΠΑ. Νομίζω ότι τώρα έχουμε περισσότερα περιθώρια, είναι πιο εύκολη η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. σκέψει σκέψεις έχω. Σύντομες. Πρώτα-πρώτα να τάξουμε ω προτεραιότητά μα στρατηγική του Αφγανιστάν. Θεωρώ ότι ήδη εδώ και δεκαετίε έχει τεθεί ω θέμα το ότι θα πρέπει να έχουμε μια πλατφόρμα κοινών αξιών, ε, κοινών ιδεών και επομένως θα πρέπει πάνω σε αυτό να χτίσουμε την αξιοπιστία μας ούτως ώστε να νομιμοποιηθεί η παρέμβαση και η επέμβαση στο Αφγανιστάν. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να ξεχαστούν κάποια θεματάκια. Για παράδειγμα, τι γίνεται όσον αφορά τις επιχειρήσεις επιτόπου. Ε, τι ακριβώς θα κάνουμε εκεί. Μας προβληματίζει πάρα πολύ βαθιά το ότι εκεί έχουμε πάρα πολλές απώλειες από τον άμαχο πληθυσμό πολιτών. Άρα θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη συνεργασία ούτως ώστε να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής, την, την, την καθημερινή πραγματικότητα των Αφγανών. Αυτό πρέπει να γίνει για τον άμαχο πληθυσμό. Περισσότερη προσπάθεια να τους βελτιώσουμε τον καθημερινό τους βίο. Να σταματήσουν να κινδυνεύουν και έτσι να σταματήσει να δέχεται πλήγματα και η αξιοπιστία μας. Τώρα κάτι άλλο. Την Μέση Ανατολή θέλω να αναφέρω τώρα. Γιατί στην Μέση Ανατολή έχουμε κάτι σαν ε, ε ένα, ένα, ένα οπλοστάσιο της τρομοκρατίας. Εκεί γεννιούνται τρομοκράτε, Βλέπουμε τι γίνεται εκεί Πόσοι νέοι στρέφονται προς ε, αυτή την κατεύθυνση λόγω των όσων γίνονται εκεί. Επομένω, όπω το έχουμε πει και στο παρελθόν, θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε τι θα γίνει με την Μέση Ανατολή και αυτό να μα προβληματίσει βαθιά. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η πρόεδρο. Και τώρα, ο κύριο Μακτσέν από το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει τώρα το λόγο. Θα σε ευχαριστώ, διότι να θέλω να σα αναφέρω. Πρώτον, ενότητα ή κοινή οπτική γωνία των μεν και των δε. Είπα Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΝΑΤΟ ή πρώτα πρώτα θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε πώς θα έχουμε κοινή οπτική των πραγματών εδώ, στα, στους κόλπους Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει υπάρχει κοινό όραμα, κοινή άποψη των πραγμάτων, γιατί έστειλε 20.000 ε, στρατιώτες, 2.000 ε, τεθωρακισμένα, κινητοποίησε η Ρωσία την αεροπορία για το ναυτικό για να επιτευχθεί στην ε, Γεωργία. Όχι, δεν ήταν ένα χωριουδάκι. Ήταν μια τεράστια κλίμακα η εισβολή που έλαβε χώρα, η πιο μεγάλη από το 1939. Κάναμε τίποτα, αντιδράσαμε. μα πήρε κάτι, κάτι εβδομάδες, κάνα μήνα για να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή γραμμή. Κάναμε τίποτα, βρήκαμε επομένω αυτό το κοινή γραμμή. Όχι, είναι απάντηση. Επομένω θα πρέπει να βρεθεί και ένα παρονομαστή στην εξωτερική πολιτική. Ιδάλω είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάτσουμε και να μιλήσουμε με του Αμερικάνου και να του πούμε συμφωνήστε μαζί μα όταν εμεί μεταξύ μα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν υπάρχει το εμεί με, με άλλα λόγια. Επίση, φυσικά και συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή ότι θα πρέπει να ε, ε, ε, συμφωνώ σε, επίπεδο ορολογίας με αυτόν τον παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Όμως, όμως για να δούμε μια, να μια ματιά στην φρασιολογία την χθεσινή. Δεν λέγαμε τότε global war, terrorism, δεν λέγαμε παγκόσμιος πόλεμος. Ε, αυτό το χρησιμοποίησαν εκείνοι. Εκείνοι έχουν κηρύξει παγκόσμιο πόλεμο εναντίον μα και πολλοί συνάδελφοι σε αυτή την αίθουσα ίσως δεν, δεν, δεν ε, παίζουν κρίκετ, δεν ξέρουν κρίκετ. Παίζεται αργά-αργά, κρατάει ένα μάτς πέντε μέρες, είναι περίεργοι κανόνες και ε, τελικά ο στόχος είναι η ισοπαλία και όχι η νίκη που κανένας από το τένις και από το πόσο και από το μπάσκετ δεν τα ξέρει αυτά. Τι έγινε τώρα. Το Πακιστάν πλέον δεν είναι δύναμη στο κρίκετ. Παρ' παρόλα αυτά όμως μπορεί να δει εκεί πέρα στο Πακιστάν και στην Κεϊλάνια ε, σε κάθε γειτονιά, παιδάκια να παίζουν, ε, του φαίνεται σαν παστικό. Επομένω, τι γίνεται τώρα. Οι τρομοκράτε τι κάνανε, δεν επιτέθηκαν σε κανένα Υπουργείο. Ε, προσπάθησαν να θίξουν αυτό να πάρουν το Πακιστάν αυτή το, το, το, κομμάτι της ταυτότητα πολιτικής. Δηλαδή να στερήσουν τους Πακιστανούς την ευχαρίστηση του κρίκετ. Εμεί έχουμε καμία στρατηγική για να βοηθήσουμε το Πακιστάν σε αυτό το επίπεδο. Διότι όπω ξέρετε οι Ταλιμπάν τώρα φεύγουν από το Αφγανιστάν και πάνε στο Καράτσε. Φεύγουν από τα στρατόπεδα, πάνε εκεί. Και η Ινδία εκεί έχει 500 εκατομμύρια στρατιώτε. πολύ πρόσφατο από όλο το ΝΑΤΟ. Έχουμε 70.000 μουσουλμάνους που έχουν σκοτωθεί στο Κασμίρ ε, τα τελευταία 20 χρόνια, οπότε όλος αυτός ο στρατός του Πακιστάν βρίσκεται στα δυτικά σύνορα. Θυμάσαι, Στίβεν, πήγαμε εκεί επί τόπου. Επομένως, ο στρατός του Πακιστάν είναι εκεί. Είναι περίπου όπως ήταν οι γερμανογαλλικές σχέσεις, δηλαδή που είχαν παραταχθεί στο θέμα και περιμένανε τον, τον πόλεμο, την εισβολή. Τι θα γίνει τώρα. Τι, δεν θα πρέπει να κάνουμε κάποια κίνηση στρατηγική ως προς την Ινδία. Τώρα, για να καταλήξω, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στον ΝΑΤΟ θα πρέπει να ε, καταλάβουμε ότι έχει αυτό το τίμημά του. Δεν μπορώ να ανήκω σε μια λέσχη άμα δεν πληρώνω συνδρομή. Το 2% του ΑΕΠ που είναι το μισό από όσο πλέον οι Αμερικανοί, θα πρέπει να είναι το ελάχιστο, η ελάχιστη συνδρομή στη λέσχη αυτή στο ΝΑΤΟ. Αν κάνει δεν θέλει να καταλάβει αυτά τα λεφτά, ωραία, ας ε, το, το παραδεχτεί, δάλο ε, να μην μένει στα λόγια, αλλά να προχωρήσει σε έργα. Η πρόεδρο. Άνικη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δόκτωρα Χάμιλτον δεν βλέπω το όνομά σα από εδώ, ζητώ συγγνώμη λέει πρόεδρος. Η παρουσίαση του κυρίου Χάμιλτον είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν και βάζει πάρα πολλά ερωτηματικά και δημιουργεί πολλές απορίες, απορίες τις οποίες θα ήθελα να μπορέσω να σας παρουσιάσω μέσα σε δύο λεπτά. Πρώτον, μου άρεσε πάρα πολύ κύριε Χάμιλτον το ότι αναφέρεστε στις σχέσεις ανάμεσα στις, Ευρωπαϊκές, ε, στις και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές και το ΝΑΤΟ στην ουσία φέρνει σε επαφή του πρωταγωνιστές τη ε, Βορειοατλαντική σχέση. Ευχαριστώ λοιπόν που αναφέρεστε στις σχέσεις ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ένωση. Και οδηγούμε τώρα στην εξή ερώτηση. Πιστεύετε πράγματι ότι πράγματι υπάρχει μια αλλαγή στη Ουάσιγκτον, την βιώνουμε την αλλαγή αυτή. Ακούσαμε και τη δήλωση του γερουσιαστή Biden. Πιστεύετε πως πηγαίνουμε όμως σε μια αλλαγή σε βάθος που θα αντικαταστήσει το αμερικανικό leadership από ένα ευρωπαϊκό partnership ανάμεσα στην Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Αυτό είναι το κλειδί και είναι και η επιθυμία της Γαλλίας. Και η επιστροφή της Γαλλίας, την οποία εγώ χειροκροτώ προσωπικά, οι περισσότεροι χειροκροτούμε προσωπικά, αλλά βέβαια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για πολιτικούς λόγους είναι εναντίον της επιστροφής της Γαλλίας στο στρατιωτικό τμήμα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει η δυνατότητα εκ νέου να οικοδομήσουμε μια σχέση ανάμεσα στην Ένωση και τη ΣΥΠΑ σωστή. Μια άλλη ερώτηση. Θα πρέπει, όπως είπατε άλλωστε, να διαμορφώσουμε ένα νέο στρατηγικό ε, σύστημα σκέψης. Και αναφέρομαι εδώ στο τι θα γίνει στις σχέσεις με τη Ρωσία. Ποτέ δεν θα οικοδομήσουμε μια πραγματική ασφάλεια στην Ευρώπη εκτός Ρωσίας, χωρίς τη Ρωσία. Και εμένατε σε αυτό και θα ήθελα να επανέλθετε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες τις οποίες θα πρέπει να πάρουμε ε, προς τη Ρωσία έτσι ώστε να την αγκυρώσουμε στην βορειοατλαντική σχέση και σε συνεργασία και με τη συνάδελφο Ριγιάκ ε, μας εξέπληξε λίγο αυτό το οποίο είπατε για τις προτινόμενες αλλαγές στον τομέα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για την επανένταξη της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ αυτός ο κανόνας, ο κανόνας της συνένεσης είναι ένας κανόνας ο οποίος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να φυγεί. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η μία ήδη έχει τεθεί από τον κύριο Μπουβάρ. Για τη Ρωσία Εμείς ε, ακούσαμε διάφορες απόψεις της Αμερικανικής κυβέρνησης ε, και ακούσαμε και για επιστολές προς τη Ρωσία σε σχέση με την πυραυλική άμυνα και κάτι το οποίο θα ήθελα να σχολιάσετε λίγο περισσότερο. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα στις Ηνωμένε Πολιτείες σχετικά με το δόγμα της πυρηνικής αποτροπής του ΝΑΤΟ και τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι θα υπάρξουν για το δόγμα αυτό και από πλευράς των ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες είναι πυρηνικές δυνάμεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Ίσως λίγο ασυντόνιστα. Με το Ιράν θα ξεκινήσω γιατί αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Εγώ μιλάω σε προσωπική βάση, έτσι δεν είναι, δεν εκπροσωπώ κανέναν, είναι σαφές αυτό, δεν εκπροσωπώ σε καμία περίπτωση κάποια επίσημη άποψη. Θα έλεγα όμως ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να δει το Ιράν με διαφορετικό τρόπο. Ελπίζω ότι ο σκεπτικισμός μας να μην βασιστεί σε παλιότερες αντιλήψεις και να μην μιλάμε συνεχώς για κυρώσεις. Η νέα κυβέρνηση είπε ότι θα περάσει σε άμεσες συζητήσεις με το Ιράν. Η προσπάθεια λοιπόν που γίνεται τώρα είναι αντίθετη με τη λογική των κυρώσεων. Τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με την πρόταση αυτή. Οι Ευρωπαίοι φίλοι οι οποίοι πιέζουν τις ΗΠΑ να έρθουν σε επαφή με το Ιράν τώρα είναι λίγο ανήσυχοι γιατί σου λέει τι θα συζητήσουν οι Αμερικανοί με τους Πέρσες. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες από πλευρά της Ευρώπης και στο τέλος αυτά που θέλει τεχεράν η Ευρώπη δεν μπορεί να τις τα δώσει. Δηλαδή μια διαφορετική σχέση ασφαλείας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θέλουμε εμείς τη ΣΥΠΑ δηλαδή να συζητήσουμε πολλά πράγματα με το Ιράν, όχι μόνο για τους βαλιστικούς πυράβλους, όχι μόνο για την πυρηνική, τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, αλλά γενικότερα για την κατάσταση στην περιοχή. Πιστεύω λοιπόν ότι η Αμερικανική κυβέρνηση είναι σαφέστατα δεκτική για τον διάλογο αυτό με το Ιράν Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι ο διάλογος μπορεί να προχωρήσει μέχρι σε ένα σημείο. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η κατάληξη και ο άλλος δρόμος, ο σκληρός θα έλεγα και αυτός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος. Θα πρέπει να έχουμε ένα καλό διάλογο με την Τεχεράνη και θα είναι καλός ο διάλογος αυτός εφόσον κατανοήσουν οι Πέρσες ότι έχουμε και άλλες δυνατότητες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί λοιπόν και στον τομέα των κυρώσεων και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να γνωρίζουν για το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση κατά την οποία ο διάλογος αυτός δεν προχωρήσει όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν κάποια κίνητρα τα οποία μπορούμε να παρέχουμε προς το Ιράν στον τομέα της ασφάλειας, σαν παράδειγμα. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες ε, ε, στον τομέα αυτό που πράγματα μάλλον που έχουν αλλάξει. Είναι δύσκολο να πει σήμερα κανείς ότι δεν θα παράγει στο μέλλον πυρηνικά όπλα το Ιράν ή ότι η τεχνολογία των βαλιστικών ε, πυράβλων αλλά από την άλλη το Ιράν πρέπει να κάνει κάποια βασικά πράγματα όπως να αναγνωρίσει την ύπαρξη του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ. Και φυσικά θα πρέπει να εμπλέξουμε και άλλες σημαντικές χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας όπως η Ρωσία και η Κίνα για να προχωρήσει ο διάλογος όπως θα έπρεπε σοβαρά. Πάντως υπάρχει μια νέα όφηση και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε σε αυτή τη φάση. Για τη Ρωσία τώρα. Θα ήθελα να πω ότι Θέλω να σας ζητήσω παρακαλώ να διαβάσετε την ίδια την έκθεση γιατί η περίληψη την οποία παρουσιάζουμε είναι πολύ μα πολύ συνοπτική. Έχουμε ολόκληρο κεφάλαιο για τη Ρωσία και θα δείτε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Εμείς υποστηρίζουμε, τα επιχειρήματά μας λένε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διτή στρατηγική. Η Ρωσία η σημερινή δεν είναι η Σοβιετική Ένωση, δεν κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις πια. Αν δει την παλιότερη κανείς ιστορία όμως της περιοχής, στο παρελθόν είχαμε κάποιες επιτυχίες με τη Μόσχα, προσπαθώντας να συνδυάσουμε δύο διαφορετικά πράγματα, δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνδυάζονται. Αν οι Ρώσοι ηγέτες λέγουν και αντιμετωπίζουν πράγματι κάποια πάρα πολύ σημαντικά εσωτερικά προβλήματα στον τομέα της υγείας, στον τομέα της δημογραφίας, στον τομέα τον οικονομικό θα πρέπει δηλαδή να περάσει από μια οικονομία η οποία είναι αυτή τη στιγμή η οικονομία που βασίζεται μόνο στις, στους ε, βασικούς, στα βασικά ε, πρώτα υλικά όπως πετρέλαιο κτλ. Αν αλλάξει λοιπόν κάπως η, Ευρωπαϊκή, η Ρωσία τότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη Ρωσία να ενταχθεί και σε πάρα πολλούς διεθνείς οργανισμούς και θα γίνουμε οι βασικοί σας εταίροι να πούμε στους Ρώσους. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες λοιπόν προτάσεις στην έκθεσή μας όπου λέμε ότι εμείς θέλουμε να περάσουμε σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ελέγχου των εξοπλισμών και εδώ είμαστε ηγέτιδα δύναμη ακριβώς λόγω της φύσης των συγκεκριμένων προβλημάτων. Από πλευρά των ε, Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να απαλλαγούμε από κάποιες νομικές ρυθμίσεις του παρελθόντος οι οποίες είναι αναχρονιστικές και δεν αντικατοπτρίζουν τις οικονομικές σχέσεις που έχουμε με τη Ρωσία. Και σε σχέση με το Ιράν μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ρώσους. Έχουμε μια συμφωνία επίσης με τους Ρώσους και για το τράνζιτ μέσω του Αφγανιστάν Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε αναλυτικά στα πλαίσια μιας θετικής θα έλεγα ημερήσιας διάταξης με τους Ρώσους. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι αρχές αυτές, οι συζητήσεις συγγνώμη αυτές θα βασιστούν σε ορισμένες αρχές όπως οι αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκη που όλοι έχουμε υπογράψει. Οι αρχές αυτές αφορούν και τα εσωτερικά θέματα των χωρών που έχουν υπογράψει και όχι μόνο τα εξωτερικά και τις διμερείς σχέσεις αν η βάση, εν πάση περιπτώσει, τη συμφωνίας είναι η αποδοχή της λεγόμενης λογικής των, των, των περιφερειών επιρροής, των ζωνών επιρροής, αυτό είναι εντελώς μη παραγωγικό σαν λογική. Αν μπορέσει να προχωρήσει ο διάλογος θα πρέπει να γίνει έχοντας απαλλαγή από ορισμένα προβλήματα του παρελθόντος. Ε, θα πρέπει η Ρωσία να σεβαστεί την αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ευρώπης. Να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις των Ρώσων και να δεχθούμε κάποιες από τις προτάσεις αυτές επί τη βάση συγκεκριμένων αρχών όπως το Ελσίνκι. Δεν χρειάζεται να πάμε πιο πίσω από το Ελσίνκι. Κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε διάλογο με εμπιστοσύνη από πλευράς μας για το ποια θα πρέπει να είναι η νέα αρχιτεκτονική των σχέσεων με τη Ρωσία επί τη βάση των συγκεκριμένων βέβαια σταθερών αρχών. Αυτού του είδους ε, η αντιμετώπιση απαιτεί θα έλεγα μία σε βάθος ανάλυση των σχέσεων των στρατηγικών ανάμεσα στην Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Δεν μπορεί κανείς να τα κάνει αυτά μεμονωμένα σαν χώρα. Δεν μπορεί κανείς να ξεπουλάει τις αρχές του. Κάποιες χώρες πιστεύουν ε, ότι θα πρέπει να εμένουν στις αρχές και να μην προχωρούν σε πρακτικά βήματα, άλλες το αντίθετο. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να γίνουν εφόσον υπάρξει μια συμφωνία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΕ. Μίλησα και για τα CBT. Εδώ έχουμε μια νέα όθηση. Θα υπάρξει μια νέα όθηση για επικύρωση της συμφωνίας αυτής θα πρέπει να δει κανείς ποια είναι η δυναμική της Αμερικανικής γερουσίας σε αυτή τη φάση. Η ενέργειά μας απορροφάται κυρίως από την οικονομική κρίση. Αλλά προσπαθούμε παρόλα αυτά να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα ελέγχου της διάδοσης των όπλων και αυτό έχει άμεση σχέση και με την κοινή γνώμη των ΗΠΑ και τα θέματα της ασφάλειας γενικότερα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν κενά αυτή τη στιγμή στα επίπεδα εξουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και ενώ στην Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα κάποια επίπεδα εξουσίας να λειτουργούν. Θα απαιτηθεί χρόνος για να λειτουργήσει το σύνολο της Αμερικανικής κυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν όταν έχετε προσδοκίες να είστε λίγο επιφυλακτικοί γιατί δεν είμαστε ακόμα μια λειτουργικά μια λειτουργική κυβέρνηση για το θέμα των πυρηνικών δυνάμεων. Στην έκθεσή μας λέγουμε ότι τίποτα από αυτά τα οποία προτείνουμε εδώ δεν θα είναι αντίθετο με τις προτάσεις που οδηγούν στο λεγόμενο παγκόσμιο μηδέν, το Global Zero. Είναι πολύ καλός ο στόχος αυτός και ποιος δεν το θέλει τον στόχο αυτό. Αλλά βέβαια τα πράγματα, ε, η πραγματικότητα μάλλον σήμερα είναι διαφορετική και θα πρέπει να δούμε τι βήματα μπορούμε να πάρουμε για να οδηγηθούμε προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου. Προφανώς η ατζέντα ε, θα πρέπει, για τον έλεγχο των εξοπλισμών θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Να δούμε και ποιος είναι ο ρόλος των πυρηνικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Παναλαμβάνω εγώ λέω μεταφέρω προσωπικές απόψεις. Ο πυρήνας λοιπόν της συζήτησης ποιος είναι. Αυτά τα όπλα τα οποία υπάρχουν σήμερα, τα οποία λειτουργήσαν σαν συμβολική αποτρεπτική δύναμη που συνδέει τις Ηνωμένε Πολιτείε με την Ευρώπη, είναι μια απόδειξη θα έλεγα ε, τελική της ε, συμμετοχής και της συνδρομής των Ηνωμένων Πολιτειών στην συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης. Αν θέλουμε να απομακρύνουμε τις προτάσεις αυτές από την Ευρώπη, για να γίνει αυτό η πρόταση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Αν οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζονται την αποτρεπτική δύναμη αυτών των όπλων και ότι μπορεί να γίνει ε, διασφάλιση της ασφάλειάς τους εκτός ΗΠΑ, να μας το πείτε. Η συζήτηση δηλαδή εσείς πρέπει να την κάνετε σαν Ευρωπαίοι. Βέβαια, ορισμένοι συνάδελφοι στο Πεντάγωνο, στι Ηνωμένε Πολιτείε γενικότερα, πιστεύουν ότι εντάξει εμείς κάνουμε τις ζητέ μα συζητήσει, μια και είναι δικά μας τα όπλα εμείς θα αποφασίσουμε τι θα τα κάνουμε. Δεν το αποκλείω αυτό, εγώ δεν θα το ήθελα αυτό γιατί είναι ανυπόμονοι πολλοί Αμερικανοί και σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο συζητούν ορισμένα πράγματα οι Ευρωπαίοι. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πει με μια ενιαία φωνή ότι θα πρέπει να φύγουν τα όπλα αυτά από την Ευρώπη γιατί είμαστε επεπισμένοι και έχουμε εμπιστοσύνη ε, στην άποψη ότι δεν έχουμε ανάγκη αυτά τα όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεχθούν το μήνυμα αυτό, θα δεχθούν μια τέτοια δήλωση. Αλλά για να γίνει αυτή η κίνηση θα πρέπει να απευθυνθεί μια, ένα αίτημα αν θέλετε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη ΣΥΠΑ. Η Ευρώπη είναι κυρίαρχη και θα αποφασίσει για αυτά. Για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξαν πάρα πολλές ερωτήσεις και η βασική μας ιδέα ποια είναι, θα την επαναλάβω. Αυτό το νέο πλαίσιο σχέσεων που δημιουργήθηκε το 1995 καλύπτει τέσσερα καλάθια θα έλεγα θεμάτων και καταρχάς προσπαθούμε να κάνουμε κοινέ αξιολογήσεις φαινομένων για να οδηγηθούμε ίσως σε κοινέ δράσεις. Δεν υπάρχει στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας του 1995 υποχρέωση θα έλεγα στρατηγικής σχέσης. Μέσω του ΝΑΤΟ ναι, αλλά όχι στα πλαίσια των σε εισαγωγικά διμερών σχέσεων ήπα Ένωσης. Το θέμα λοιπόν της στρατηγικής συμμαχίας είναι ένα θέμα ανοιχτό. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να εκφράζουμε ε, αυτή την αίσθηση αλληλεγγύης που έχουμε στις σχέσεις μας. Και πώς θα το κάνουμε αυτό, πώς, τι σημαίνει αυτή η αλληλεγγύη. Δεν θέλω εγώ να, να παρέμβω στις συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρήτρα της αλληλεγγύης. Αλλά μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι απλά σύμμαχοι αλλά και στρατηγικοί εταίροι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αν υπάρξει κάποια καταστροφή ή οτιδήποτε άλλο τι θα κάνουμε. Εγώ παρακολουθώ επίσης και αυτά που λέγουν οι μη ε, συντεταγμένες πολιτικά χώρες όπως η Σουηδία και τα λοιπά ότι στην περίπτωση ε, όπου υπάρξει κάποιο πολύ σοβαρό διεθνές συμβάν θα παραμείνουν παθητικοί θα μπορούσαμε να το πούμε εμείς μεταξύ μας αυτό. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα τα πράγματα. Τα τέσσερα καλάθια των σχέσεων δεν ακαλύπτουν ορισμένους τομείς όπως η ενίσχυση της αντοχής της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Τα θέματα που συζητιούνται είναι πολλά και πρότασή μας είναι να κάνουμε μια νέα μελέτη όπως αυτή την οποία προτείνουμε για τον ΝΑΤΟ και για τις σχέσεις ανάμεσα στην Ένωση και τη ΣΥΠΑ και με κοινοβουλευτικές διαστάσεις, να συνεργαστούμε με την Τσεχική και τη Σουηδική Προεδρία, να κάνουμε προτάσεις και προς την Ισπανική Προεδρία η οποία εν πολύ στο 1995 ήταν υπεύθυνη και για τη νέα ε, διατλαντική στρατηγική και να δούμε επί τη βάση ποιων προτάσεων θα οικοδομήσουμε αυτή τη νέα στρατηγική σχέση. Νομίζω ότι το θέμα της ενίσχυσης της αντοχής των κοινωνιών μας είναι θα έλεγα ένα κομβικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν ε, κάποια κοινωνικά προβλήματα αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια πρώτη φάση να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Ανθρωπιστική βοήθεια σαν παράδειγμα η ΕΠΑ και η Ένωση μήπως πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο. Όλα αυτά μπορούμε να τα εξετάσουμε. Έχουμε πάρα πολλές ιδέες για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Θα τα συζητήσουμε αυτό σε μια άλλη αφορμή, μια άλλη φορά. Με ρωτήσατε τι μπορούν να κάνουν οι βουλευτές της Ηνωμένε Πολιτείες για να υπάρξει περαιτέρω κατανόηση. Εγώ είμαι διευθυντής του κέντρου του Πανεπιστημιακού ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΣΥΠΑ. Εγώ είμαι ε, διευθυντής του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Κέντρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουάσιγκτον. Μπορούμε να κάνουμε κάποια, προβλη... βήματα προόδου, μελέτες, επιστοποιημένες μελέτες, κοινά μαθήματα ανάμεσα ε, σκηνή διδακτέα ύλη, ανάμεσα σε διαφορετικά αμερικανικά πανεπιστήμια της πολιτείας στη Ουάσιγκτον Υπάρχουν εκτός από το δικό μας άλλα δέκα τέτοια πανεπιστημιακά ευρωπαϊκά κέντρα. Είναι καλή αυτή η επένδυση την οποία κάνετε τη. Νομίζω λοιπόν ότι όπως είπα υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες στη σχέση μας σήμερα. Ε, ξέρετε ότι οι προτάσεις που έγιναν του 1995 ε, προτάθηκαν από διάφορα think tanks και ε, το τελευταίο καλάθι όπως λέγαμε είναι κάτι το οποίο είχε προταθεί από πανεπιστημιακούς και ήταν λίγο θεωρητικό. Αυτό το οποίο προτείνουμε για το τέταρτο καλάθι δεν έχει την απόλυτα κοινοβουλευτική διάσταση την οποία θα θέλαμε. Ακόμα και αν οι δημοκράτες τότε ήταν πλειοψηφία, είχαν τις δικές τους προτεραιότητες και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες νέες ρυθμίσεις έτσι ώστε η κοινοβουλευτική διάσταση της συνεργασίας είπα Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανεξεταστεί. Να εξεταστεί εκ νέου λοιπόν από κοινού και αυτό είναι μια κοινή προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Ο Τούρκος συνάδελφος είπε για τον τρόπο λειτουργίας τις σχέσεις αυτές. Εγώ δεν προτείνω αυτή τη στιγμή μια πλήρη αναδόμηση των σχέσεων μέσα στο ΝΑΤΟ. Προφανώς και το ΝΑΤΟ είναι ο κεντρικός χώρος συνεργασίας στα θέματα ασφαλείας και πρέπει να παραμείνει σαν τέτοιος. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα στα οποία συνεργαζόμαστε. Η διαδικασία της ομάδας των 20, το G20 σαν παράδειγμα. Προφανώς ο πυρήνας αυτής της προσπάθειας όπως είπα είναι καθοριστικός και είναι διατλαντικός, όχι απαρκής από μόνος του βέβαια το πώς θα, γίνουν, θα λαμβάνονται αποφάσεις, το πώς ε, θα σταθμίζονται οι αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, ε, σίγουρα από μόνη της η διατλαντική διάσταση δεν αρκεί. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τη χρηστή διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι υπάρχουν νέες δυνάμεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά δεν συμμερίζονται τις ίδιες αρχές με μας. Θα πρέπει να το συζητήσουμε λίγο και το θέμα αυτό. Εμείς μερικές φορές δεν σταθήκαμε και στο ύψος των υποσχέσεών μας, αλλά παρόλα αυτά τηρήσαμε την βάση των προσδοκιών των πληθυσμών, δηλαδή οι αρχές της μη διάκρισης, η σωστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και εμείς θα πρέπει να είμαστε από τους βασικούς πρωταγωνιστές μιας τέτοιας συζήτησης. Επανέρχομαι στα θέματα της ενίσχυσης της αντοχής των δύο εταίρων. Από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς που δημιουργήσαμε τον τελευταίο καιρό για να αντιμετωπίσουμε μη ορθόδοξες επιθέσεις είναι οι νέες μορφές διεθνών ομαδοποιήσεων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Κάποιες είναι καρπός της συνεργασίας της ομάδας των 8, η ομάδα ας πούμε δράσης στον τομέα των, χρηματοπιστωτικών δημιουργήθηκε ήδη από το 1999 για να εξετάσει τα θέματα της διακυβέρνησης της οικονομίας. Η ομάδα της Λιών ε, δεν είναι επίσημες οι δομές αυτές, δεν είναι θεσμική αν θέλετε η δημιουργία τους. Παρ' όλα αυτά ασχολούνται με αρκετά θέματα. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέα δίκτυα, πρέπει να δημιουργήσουμε τα δικά μας δίκτυα, τα οποία πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα, ελαστικά. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες διαβούλευσης και βελτίωσης της διαβούλευσης και για την Τουρκία. Ίσως θα πρέπει να βρούμε και περιφερειακούς τρόπους συνεργασίας. Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχει καταστεί για μας μείζον στρατηγική περιοχή. Η Τουρκία έχει προτείνει ένα σχέδιο, ένα σύμφωνο ε, σταθερότητας του Καυκάσου, εν πάση περιπτώσει, ή κάτι τέτοιο. Ε, ήμουνα κάποτε υπεύθυνο για το σύμφωνο σταθερότητας και έχω κολλήσει σε τέτοιες ε, ορολογίες. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι μια νέα μορφή δικτύου, είναι νέες ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν σε επαφή εντελώς διαφορετικούς πρωταγωνιστές που προέρχονται από την Ευρώπη και πέραν της Ευρώπης. Να δημιουργήσουμε δηλαδή νέες ε, δυνατότητες για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα αλλά να μπορούν να γίνουν στο μέλλον. Μιλάμε για μια περιοχή, θυμίζω τον Κάφκασο, η οποία είναι ελαφρώς ασταθής. Πρέπει να βοηθήσουμε τους πληθυσμούς να δούνε ε, πού είναι το μέλλον τους. Το ίδιο είχαμε να κάνουμε και στα Βαλκάνια πριν αρκετά χρόνια. Τότε ήταν και τμήμα της Ευρώπης και είναι τμήμα φυσικά της Ευρώπης, αλλά και εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα. Ευτυχώς όμως αποφασίσαμε να πούμε ότι μπορείτε να έρθετε εδώ που είμαστε εμείς, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό, να μπουν στην Ένωση δηλαδή. Να μην μιλάμε δηλαδή μόνο για θεσμικά, αλλά να μιλάμε για την ουσία, για τις προϋποθέσεις. Μπας μου ζητάνε να κλείσω Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, δεν ξέρω τι έχω αφήσει, χωρίς να θέλω να παραβιάσω την προσταγή της Προέδρου. Ένα θέμα το οποίο επανέρχεται συνεχώς για συζήτηση είναι το Αφγανιστάν. Επαναλαμβάνω λοιπόν για το Αφγανιστάν. Οι κίνδυνοι που προέρχονται από τα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν είναι η πιο οξία και άμεση απειλή για τους Βορειοαμερικανούς και τους Ευρωπαίους σήμερα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη φύση του κινδύνου αυτού, τη συγκεκριμένη πρόκληση, και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τη σοβαρότητα που του αξίζει. Το θέμα δεν είναι μόνο να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία στο Αφγανιστάν. Το θέμα είναι να εξορκίσουμε την τρομοκρατία από το σύνολο αυτής της περιοχής για να μην θίγει τους πληθυσμούς. Αυτός είναι ο στόχος. Περιορισμένος είναι μάλλον ο στόχος. Αλλά για να τον πετύχουμε τον συγκεκριμένο στόχο πολλά θα πρέπει να γίνουν και όχι μόνο στον στρατιωτικό τομέα, στον τομέα της πολιτικής διακυβέρνησης, στον τομέα της οικονομίας και αυτό άπτεται και του Πακιστάν. Οπότε ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Πακιστάν. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Αν πρέπει να συνεργαστούμε, αν πραγματικά θέλουμε να παίξουμε ένα κεντρικό διεθνή ρόλο, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν έχω ακούσει τίποτα για τη στρατηγική της Ένωσης προς το Αφγανιστάν και για τη σταθεροποίηση της χώρας. Και τι κάνει εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με το Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ δεν θα μπορέσει να πετύχει εάν δεν υποστηρίζεται στις προσπάθειές του από άλλους εταίρους. Ακόμα και η συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών θα έλεγα θα πρέπει να ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο. Στα γερμανικά συνεχίζει. Ε, προς τον Γερμανό ε, Ευρωβουλευτή, οι, οι λεγόμενες home missions, συνεχίζει τα αγγλικά ε, όταν λέω home missions εννοώ βεβαίως την επικράτεια των χωρών που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ. Βέβαια για 50 χρόνια κυρίως ήταν η Γερμανία και οι περισσότεροι Γερμανοί νομίζω τότε θεωρούσαν ότι το ΝΑΤΟ προστατεύει την Γερμανία. Ότι η αποστολή του ΝΑΤΟ καθαρά ήταν home mission. Οι Γερμανοί τώρα βέβαια καλούνται να βγουν να πάνε να προστατεύσουν άλλους. Αυτό είναι η μεγάλη συζήτηση που γίνεται στη Γερμανία και μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αλλά ε, home missions νομίζω ότι είναι μια έννοια που γνωρίζουν οι Γερμανοί διότι το ΝΑΤΟ επέτυχε ακριβώς επειδή είχε δεσμευτεί να κάνει home mission. Ε, ίσως είναι θέμα ορολογίας. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της ανθεκτικότητας των κοινωνιών, διαβάστε την έκθεση επειδή πολλοί ρωτήσατε σχετικά. Εμείς δεν λέμε να μπει ο στρατός σε θέματα μη στρατιωτικά. Δεν λέμε να παραβιαστούν κάποιες βασικές αρχές που όλοι γνωρίζουμε. Λέμε ότι η βασική σχέση θα είναι Ηνωμένε Πολιτείε και Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορα διμερεί. εμεί εξετάσαμε την ατζέντα αυτή και είδαμε σε συγκεκριμένου ρόλου το ΝΑΤΟ μπορεί να παίξει υποστηρικτικό ρόλο για την ε, ενίσχυση τη ανθεκτικότητα των, κινητών, των κοινωνιών. Χωρί βεβαίω να παραβιάζουν οι βασικέ αρχέ και κρατώντα το στρατιωτικό μέρο εκεί όπου ανήκει, στο στρατιωτικό μέρο. Δεν είναι θέμα αυτό για μας να μπουν δηλαδή οι στρατιωτικοί σε τομείς μη στρατιωτικούς. Ευχαριστώ. Ε, well, ε, it was a very interesting ε, Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση της εκθέσεώς σας. Όντως νομίζω ότι πρέπει να την διαβάσουν όλοι γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Έχοντας ακούσει λοιπόν σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που ανοίγει η νέα πολιτική των ΗΠΑ αλλά και οι προσδοκίες που έχει απέναντι στους συμμάχους της η νέα Αμερικανική κυβέρνηση θα έρθουμε σε μια ευρωπαϊκή προοπτική για το μέλλον των ε, διατλαντικών σχέσεων ασφάλειας. Έχουμε έναν άλλο λοιπόν αναγνωρισμένης αξίας ομιλητή τον κύριο Ζαβορόφσκι που είναι Research Fellow στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας στο Παρίσι και εκεί ασχολείται με τις σχέσεις με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με την εξωτερική πολιτική, με την διεύρυνση της Ένωσης και με την Ανατολική Ασία. Έχει κάνει δημοσιεύσεις για όλα αυτά τα θέματα. Προερχόμενος από την Πολωνία, ο κύριος Ζαμπορόφσκι πήρε το μάστερ σε διεθνείς σχέσεις και το έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιχαμ. Πριν να μπει στο κέντρο όπου εργάζεται τώρα το 2005 ήταν λέκτορ διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Άστον. Από το 2002 έως το 2004 ήταν και συντονιστής διατρατικών προγραμμάτων στο κέντρο αυτό για τις διεθνείς σχέσεις στη Βαρσοβία. Ο κύριος Ζαμπορόφσκι είναι και πρώην Research Fellow του ΝΑΤΟ και επισκέπτης καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Σας δίνουμε το λόγο για 10 λεπτά. Περίπου, εν πάση περιπτώσει, μετά θα ακούσετε ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι ε, μεγάλη τιμή και για μένα και για το Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι που μου επιτρέπετε να σας ομιλήσω εδώ και σε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και ελπίζω να ε, γίνει και προηγούμενο για το μέλλον. Θα προσπαθήσω να διατηρήσω τα, το χρόνο των 10 λεπτών όπως μπορώ καλύτερα και όπως έκανε και ο Ντάν θα βασίσω και εγώ την παρουσίασή μου σε μια έκθεση που έχει ε, δημοσιεύσει το Ινστιτούτο μου και από ό,τι μαθαίνω έχει διανεμηθεί σε ορισμένα μέλη. Εγώ δεν έφερα βέβαια αριθμό ε, αντιτύπων επαρκή, αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Η μελέτη μας είναι διαφορετική από την έκθεση του Νταν Χάμιλτον σε πολλές πτυχές. Αποτελεί το έργο του Ινστιτούτου μας. Άρα ε, τα όσα περιλαμβάνονται έχουν παραχθεί από τους διάφορους μελετητές που συνεργάζονται από διάφορες χώρες μέλη της Ένωσης με στόχο να ε, συντάξουμε εδώ μια ευρωπαϊκή απάντηση συντονισμένη στο Ινστιτούτο μας ε, για να εξηγήσουμε ποιες θεωρούμε ότι είναι οι βασικές προτεραιότητες στην ατζέντα των διατατικών σχέσεων για τα επόμενα χρόνια μετά από την εκλογή του νέου Πρόεδρου Ομπάμα. Εμείς αυτοπεριοριστήκαμε κατά κάποιο τρόπο στο να σημειώσουμε τις πραγματικά ε, σημαντικότερες προτεραιότητες και για την Ένωση και για τις Ενωμένες Πολιτείες. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πολύ 7 θα πρέπει να είναι αυτές και θα πρέπει να καλύψουν και την παγκόσμια ατζέντα αλλά και τις περιφερειακές. Τα Αυτά είναι η ε, Global Governance, αλλαγή του κλίματος, μη διασπορά, Ιράν, Αφγανιστάν, Ρωσία, Μέση Ανατολή και περιλαμβάνουμε και ορισμένα σχόλια σχετικά με την μεταρρύθμιση των ε, ρυθμίσεων των διατλαντικών σχέσεων. Δεν έχω βέβαια αρκετό χρόνο με 10 λεπτά για να σας τα εξηγήσω όλα αυτά. Ώστε αποφάσισα να περιοριστώ σε τρεις μόνο από αφοπλισμό και μη διασπορά, Αφγανιστάν και διατατικές ρυθμίσεις. Έρχομαι στο πρώτο. Μη διασπορά και αφοπλισμός. Αυτό το θέμα θα συζητηθεί και μετά από, στο, επόμενο δηλαδή ε, γύρο αλλά ήδη τα έχει πει και ο Ντάν. Θεωρούμε ότι η μηδενική επιλογή ως όραμα θα υιοθετηθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση και ότι θα γίνουν σχετικά βήματα. Αναμένουμε ότι θα γίνουν τρία πρώτα βήματα. Πρώτα μία δήλωση ότι ο στόχος δηλαδή της διατήρησης πυρηνικών όπλων από πλευράς ΗΠΑ είναι η αποτροπή. Δεύτερο, ότι θα γίνει μία σοβαρή προσπάθεια την ε, διάσκεψη αναθεώρησης της συνθήκης μη διασποράς το 2010 για να ενισχυθεί αυτή και, ότι θα γίνει προσπάθεια μαζί με τους Ρώσους και άλλες ε, περιφερειακές δυνάμεις να μειωθούν τα πυρηνικά όπλα σε όχι παραπάνω από χίλιες κεφαλές ανά χώρα. Και τέλος, Αυτό ε, ε, θα γίνει εάν ο Ομπάμα είναι τυχερός και εκλεγεί για δεύτερη φορά προς το τέλος μιας δεύτερης ε, θητείας του ένα βήμα δηλαδή ακόμα προς μια πλήρη κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Αυτά ίσως σας φαίνονται εντελώς φανταστικά για την ώρα. Όμως εμείς θεωρούμε ότι μια τέτοια προοπτική πράγματι θα ακολουθηθεί και από συγκεκριμένες πολιτικές. Θα έχει, θα έχει βέβαια σημαντικές επιπτώσεις, πολύ σημαντικές για την Ευρώπη. Δεν είμαι βέβαιος ότι για την ώρα γνωρίζουμε πλήρως τι έκταση παίρνει η συζήτηση αυτή στις ΗΠΑ και ότι έχουμε τις απαραίτητες απαντήσεις. Θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις χώρες που διαθέτουν πυρηνικό εξοπλισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το καθεστώς τους. Θα έχει επιπτώσεις για τις πυρηνικές δυνάμεις των Αμερικανών που είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη. Ασφαλώς θα έχει και επιπτώσεις για ορισμένες ε, χώρες της κεντρικής Ευρώπης οι οποίες εξαρτώνται πάρα πολύ για την προστασία τους από την εφιστάμενη αντιπυρηνική ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν ξέρω κατά πόσον οι κυβερνήσεις αυτές θα αντιδράσουν με ενθουσιώδη τρόπο. Βέβαια γνωρίζουμε ότι η κοινή γνώμη είναι καταρχήν ε, λίαν υπέρ ε, της ε, προσπάθειας αφοπλισμού. Δεν ξέρω βέβαια εάν οι κυβερνήσεις θα ανταποκριθούν και ίσως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι που ο Ντάν ήδη ανέφερε προηγουμένως ότι το Πεντάγωνο δηλαδή πολύ πιθανόν θα προχωρήσει στον δρόμο εφαρμογής ορισμένων πολιτικών όχι απαραίτητα ανταποκρινόμενο στις δικές μας ιδέες. Εγώ νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Το δεύτερο θέμα που επιθυμώ να σας αναπτύξω είναι το Αφγανιστάν, το οποίο και αυτό συζητήθηκε ήδη και το οποίο θα συζητηθεί ξανά και ξανά σε διάφορες περιπτώσεις. Εγώ το Αφγανιστάν το θεωρώ απολύτως πρώτη στην προτεραιότητα για τις διατρατικές σχέσεις για τα επόμενα χρόνια. Δεν θα εξαφανιστεί το θέμα αυτό. Θα παραμείνει στην ημερήσια διάταξη κάθε συζήτησης και συνάντησης με την Αμερικανική πλευρά. Η σημασία του θέματος μεγαλώνει διαρκώς. Και νομίζω ότι με τις φωνές που ακούμε καμιά φορά ε, στην Ευρώπη ότι εν πάση περιπτώσει αυτό είναι σημάδι των καιρών, θα περάσει, είναι προσωρινό, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτά είναι ευχολόγια ορισμένων και ε, θα συνεχίσει να αποτελεί ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας. Υπάρχουν σαφείς προσδοκίες από πλευράς Αμερικανών σχετικά με το ότι οι Ευρωπαίοι θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει και θα ε, συνεισφέρουν σημαντικά στην υπόθεση του Αφγανιστάν. Υπάρχει ήδη κάποια καταρχήν συνένεση ε, ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά αυτό, αυτή δεν έχει πάρει ακόμα στρατιωτική μορφή. δεν έχουμε αυξήσει τις δυνάμεις από πλευράς Ευρώπης που συμμετέχουν ε, στην ISAF στο Αφγανιστάν. Ίσως μέχρι αριθμό χιλίων ε, στρατιωτικών από όλες συνολικά τις χώρες της Ευρώπης οι οποίες ε, συμμετέχουν εκεί. Ενώ οι Αμερικανοί προτίθεται να στείλουν 30.000 πρόσθετους στρατιωτικούς εκεί. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι ο πρόεδρος Ομπάμα στην διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ δεν θα ζητήσει περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις από τους Ευρωπαίους γιατί το ξέρει ήδη ότι δεν πρόκειται να τις πάρει. Νομίζω ότι ε, τα έχουν καταλάβει αυτά οι Αμερικανοί. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προσδοκίες οι οποίες θα τεθούν και μάλιστα και με εναλλακτικέ επιλογές πώς μπορούν να βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι δηλαδή με άλλους τρόπους πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, για παράδειγμα, για την θέσπιση του κράτους δικαίου, για τη χρηστή διοίκηση, για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη στη χώρα αυτή. Ίσως πιο συγκεκριμένα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας, για την παρατήρηση εκλογών, για την εκπαίδευση δικαστών. Και επίσης αν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει πράγματι πολιτική βούληση στην Ευρώπη για να αρθούμε στο ύψος των προσδοκιών αυτών. Η αστυνομική μας αποστολή στο Αφγανιστάν δεν απέτελεσε επιτυχία και το λέω διπλωματικά. Δεν αποδίδουμε, δεν τηρούμε τα υπεσχημένα για την μεταρρύθμιση της αστυνομίας στο Αφγανιστάν. Και πολλοί μας επικρίνουν από την άλλη πλευρά του γιατί μας υπενθυμίζουν ότι υποσχεθήκαμε πριν από 8 χρόνια στην Βόνη να το πράξουμε. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στην υπόθεση του Αφγανιστάν, εμείς εδώ στην Ευρώπη πρέπει να προτείνουμε μια σοβαρή και θετική στρατηγική. Αυτά που βλέπω εγώ είναι μάλλον μια χλιαρή διάθεση σε ορισμένους ε, κύκλους εδώ σχετικά με και, και μάλλον μια διάθεση να πούμε ότι ό,τι χάσαμε χάσαμε και σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το Αφγανιστάν. Αυτό όμως θα σημάνει μια πάρα πολύ ε, σημαντική υποβάθμιση των σχέσεων με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα καταστρέψει αυτό το ε, άνοιγμα, αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή με την νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό και να είμαστε σοβαροί σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν. Το τρίτο θέμα που θα ήθελα να σας αναπτύξω είναι η ε, αναμόρφωση των διατλαντικών ρυθμίσεων. Μιλήσαμε ήδη για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ένωσης που έχουν βελτιωθεί για δύο λόγους. Πρώτον, διότι στη δεύτερη Προεδρία Μπούς η συνολικότερη αντιμετώπιση απέναντι στην Αμερικανική συγγνώμη, απέναντι στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλεια και άμυνας βελτιώθηκε σημαντικά. Κάτι το οποίο δεν πιστώνουμε πάντοτε στον πρόεδρο Μπούς και όμως είναι αλήθεια. Δεύτερο, η σχεδιαζόμενη ε, επιστροφή των Γάλλων στο στρατιωτικό σκέλος, κάτι που ε, είναι πάρα πολύ θετικό και όλοι το κρίνουν ως πολύ θετικό, έχουμε και ένα συνεχιζόμενο θέμα του εμποδίου των ε, σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας και αυτό εξακολουθεί να ανακόπτει κάθε ενδεχόμενο πρόοδου. Όμως, όπως Ακούσαμε και όπως νομίζω ότι θα συμφωνήσετε οι περισσότεροι εξημών εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΕΠ Πολιτείες μπορεί να βρεθεί τρόπος. Όχι απαραίτητα για να ξεπεραστεί πλευρικά αυτό το βασικό εμπόδιο αλλά για να βρεθούν πρακτικές ρυθμίσεις όπως για παράδειγμα κάναμε στο Κόσοβο. χωρίς να είναι ίσως απαραίτητο να προβάλλουμε ε, διαρκώς κάποια δικαιολογία, να λέμε δηλαδή ότι δεν προχωρούμε διότι υπάρχει αυτό το εμπόδιο και διότι δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο να το επιλύσουμε. Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάποια ρεαλιστικά πραγματικά μέτρα τα οποία να μπορούν να εφαρμοστούν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα εδώ είναι η διμερής σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενωμένων Πολιτειών. Βρισκόμαστε νομίζω στο σωστό χρονικό σημείο για να σκεφτούμε την ενδεχόμενη αναδιάρθρωση των υφιστάμενων σχέσεων. Για τη συνεργασία στο διμερές πλαίσιο. Εδώ αναπτύσσονται και αναφύονται πολλά θέματα. Το Ιράν εντάσσεται εδώ. Το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος. Ορισμένα θέματα του Αφγανιστάν. Η διμερής λοιπόν ατζέντα του Ατλαντικού είναι μεγάλη και όλο και μεγαλώνει. Το γεγονός ότι, ότι διεξάγονται και αιτήσεις διασκέψεις κορυφής ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα που τίθενται. Και όπως γνωρίζετε επίσης, οι διασκέψεις κορυφής δεν είναι και καλά διαρθρωμένες ώστε να εξασφαλίζουν επιτυχία. Άρα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι ορισμένες προτάσεις πρέπει να εκπονηθούν και να είναι έτοιμες ήδη για τον Απρίλιο για τη συνάντηση του Πρόεδρου Ομπάμα με τους Ευρωπαίους εδώ. Και αν όχι, τότε οι Αμερικανοί ίσως πρέπει να καταστήσουν σαφές στον Πρόεδρο Ομπάμα ότι χρειάζεται να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς θα αναδιαρθρώσουμε τις ε, σχέσεις αυτές. Το οποίο με φέρνει σε ορισμένα από τα θέματα που ε, έθεσαν οι προηγούμενοι ομιλητές είναι αλήθεια ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος ότι η σχέση αυτή δεν λειτουργεί και δεν θεσμοποιείται και αν δεν γίνει αυτό δηλαδή, ίσως οι Ηνωμένε Πολιτείε τελικώς να αποφασίσουν να μιλούν με επιλεγμένες χώρες μέλη. Και υπάρχει μια τέτοια τάση. Να πει κάποια ιεραρχία δηλαδή στους συνομιλητές από πλευρά Ευρωπαϊκής. Αυτό θα σημαίνει πολύ απλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μιλούν στις τρεις μεγάλες χώρες και αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα αποβεί σε βάρος όλων των υπολείπων. Ίσως εδώ ε, θα πρέπει να σταματήσω κυρία Πρόεδρε. Oh, uh, thank you very much. σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στη συμπρόεδρο στην Άννα Μαρία Γκόμες στη φίλη. Εγώ θα ήθελα πρώτα πρώτα να απαντήσω σε αυτό το τελευταίο το οποίο αναφέρεται. Δηλαδή πώς μπορούμε να αλλάξουμε ε, την δομή των διμερών αυτών σχέσεων με τις ε, ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να γίνει με κοινοβουλευτικές επαφές και επίσης θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τις δυνατότητες που υπάρχουν με ε, τηλεσυνεδριάσεις. ακριβώς για ασφάλεια, για άμυνα. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με συναδέλφους, έτσι, με τηλεσυνεδρίαση. Και έτσι μπορούμε να αποφύγουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Να το εξετάσουμε, να συνεργαστούμε επ' αυτού και να δούμε και κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία ε, μπορούν να μας οδηγήσουν στο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για το Αφγανιστάν τώρα. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο προσκεκλημένος μας. Ε, θεωρώ δε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι προβλήματα υπάρχουν όσον αφορά τις ε, αποστολές αυτές, τι έγινε επίσης όσον αφορά την ε, δικαιοσύνη γιατί όσον αφορά τη διακυβέρνηση εδώ έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Στο Αφγανιστάν όσον αφορά την αποκατάσταση της λειτουργίας της δικαιοσύνης και την ανοικοδόμηση της χώρας. Πάντως θα πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα μας πήγε έφυγε και μας είπε ότι σαφώς προκύπτει ότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι διαβασμένοι. Οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται για το Αφγανιστάν. Γι' αυτό και δεν περνάει το μήνυμα στον κόσμο. Μα όμως ε, πρόκειται για θέμα ασφάλειας, για θέμα άμυνας και αυτό αφορά και το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Και τώρα με τη καινούργια Αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να δούμε τι στρατηγική στροφή θα ε, σημειωθεί και από στρατηγική πλευράς, από πλευρά ανασυγκρότηση, από πλευράς ε, επαναφοράς, αποκατάστασης του κράτου δικαίου εκεί. Και να δούμε πώς τελικά θα έχουμε σοβαρή προσπάθεια και σοβαρή ευρωπαϊκή παρέμβαση. Επομένως, αυτή η πλατφόρμα συνεργασίας Ένωσης ΝΑΤΟ είναι κάτι το οποίο θα μας προσανατολίσει για τις σχέσεις μας στο μέλλον. Έχουμε, η Ένωση έχει ποτέ στρατηγία του Αφγανιστάν, δεν νομίζω. Α, ρώτησα τον κύριο Σολάνα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε. Και αν υπήρχε ήταν λάθος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο προς την κυρία Γκόμες. Ο κύριο Ονισκέδης τώρα, ε, ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριο Ονισκέδης. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε. Σε αυτή τη νέα προσέγγιση με βρίσκουν σύμφωνο. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η τάση ε, όσον αφορά το να έχουμε καλύτερη συνεργασία και έτσι και εμείς θα αναγκαστούμε να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα το τι γίνεται με την κοινή εξωτερική μας πολιτική. Δηλαδή, κάτι να μας τριμώχνεται παρά να μην κάνουμε τίποτα και απλώς να σας επικρίνουμε. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν άρτη, μια που καλούμε θα κάτι να κάνουμε από κοινό. Γι' αυτό και νομίζω ότι αυτή είναι η προσέγγιση θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλες ε, σημαντικές προσδοκίες. Τώρα, τα θέματα τα πυρηνικά. Για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την στατική των Ρώσων. Παρετήθηκαν από εκείνη τους την υπόσχεση. Δεν την τήρησαν ότι δεν θα προσφύγουν στη χρήση πυρηνικών που είχαν πει. Τώρα κατασκευάζουν εκ νέου τέτοια όπλα. Όπως πριν. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουν ε, αδυναμία μειονεκτούν όσον αφορά τις συμβατικές δυνάμεις. Άρα, δύσκολο να θεωρήσουμε ότι κάποια στιγμή θα ασπαστεί την ε, μηδενική λύση η Ρωσία. Επίσης, το Ισραήλ. για να είμαστε ξεκάθαροι το Ισραήλ έχει πυρηνικά είναι για το Ισραήλ θέμα επιβίωσης αυτό που μας να μην το ξεχνάμε αυτό άλλωστε μπήκε και στην συνθήκη για τα όπλα Έτσι, επομένω, με αυτή την οπτική γωνία νομίζω θα εξετάσουμε καλύτερα το θέμα. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριο Λαντσπέργκης τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Ζαμπορόφσκι. Ήταν ένας εκ των ε, συντακτών και συγγραφέων εκείνου του εγχειριδίου ε, το θέμα για το οποίο συζητούμε. Ρίχνω μια ματιά μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο στο κεφάλαιο 4 δεν ξέρω αν το θέμα είναι τεχνικό, τεχνοκρατικό, αλλά ίσως υπάρχει και κάποια ουσία εκεί που λέει ορισμούς, περιγραφές CIS και NIS αυτά τα, τα, τα ακρονίμια η ΚΑΚ δηλαδή, η Κοινότητα Ανεξαρτήτων Κρατών και έχουμε αυτή την ομάδα επομένως των πρώην δημοκρατιών υπό την ηγεσία της Ρωσίας και από την άλλη μεριά έχουμε τα προσφάτως ανεξαρτητοποιηθέντα κράτη. Ένα, ταυτίζονται αυτές οι δύο ομάδες κρατών ή υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Εκεί που αναφέρεται συγκεκριμένα τον χειριδιό σα στην ε, διαδικασία του μετασχηματισμού και των μεταρρυθμίσεων σε αυτές τις ομάδες κρατών. ΚΑΚ και ΕΝΑΙΕΣ και προσφάτως ανεξαρτοποιηθέντα κράτη. Ποια είναι η διαφορά. Τώρα, κάτι άλλο. Πρόκειται για αυτή την αρχή που αναφέρεται συνεχώς όσον αφορά τον χώρο τον μετασοβιετικό. Τι είναι αυτό όπως λέμε ε, η εποχή μετά την Ιγκοσλαβία η εποχή μετά την Βρετανία. Για να το ξανα Εάν το ξαναδούμε, μήπως θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η διατύπωση. Μας λέτε για αυτές τις τάσεις, ε, εθνικιστικές πολιτικές, ε, αποδημοκρατισμός εκεί στο ΚΑΚ. Η Ρωσία και αυτή είναι ΚΑΚ. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς για ε, αποδημοκρατισμό, για ε, ε, τέλος πάντων έλλειμμα δημοκρατίας ή συρρήγνωση δημοκρατίας. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί αφορούν και τη Ρωσία. Είναι συμπεράσματα από τον πόλεμο στην Γεωργία. Λέτε ότι είναι δυνατόν ή όχι να έχουμε περισσότερη ασφάλεια σε αυτό τον χώρο Είναι επιθυμία μας, γίνεται όμως σε αυτό το μετασοβιτικό χώρο. Είναι δυνατόν να υπάρχει όταν έχουμε να κάνουμε με κάποια εθνικιστική Ρωσία, δημοκρατία, συρρυκνώνεται. I'm true in such a perception or could you clarify more? Ισχύει αυτό το οποίο κατάλαβα ή όχι, μπορείτε να το διευκρινίσετε ή μήπω όσον αφορά αυτή την τάση για σύγκρουση της δημοκρατίας η μηπω οσον αφορα αυτη την ταση για συγχρονη της δημοκρατιας η ρωσια δεν συμπεριλαμβάνεται σε, σε αυτή την τάση και είναι εξαίρεση. Τι είναι, είναι τμήμα αυτού του συνόλου. Ευχαριστούμε πολύ, ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος από την Τουρκία. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι η ύψιστη προτεραιότητα το Αφγανιστάν πάρα πολλές προκλήσεις εδώ αναδύονται πρώτα πρώτα όσον αφορά την χρηστή διακυβέρνηση στο Αφγανιστάν όπου δυστυχώς η κυβέρνηση Καρζάη αποδυναμώνεται έχουμε φαινόμενα διαφθοράς οπότε και ο πόντρος στόχος μας είναι να υπάρξει μεταβίβαση της εξουσίας στην κυβέρνηση Αφγανών σε δύο, 3 χρόνια άρα χρειάζεται κάποια αξιοπιστία διότι εάν ο λαός του Αφγανιστάν απολέσει την εμπιστοσύνη, την ελπίδα, τις προσδοκίες προς την κυβέρνηση, αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό χτύπημα. Γι' αυτό είναι ερώτηση φυσικά και προς τους δύο εισηγητές μας. Υπάρχει στρατηγική. Καταβάλλονται τίποτε προσπάθειες τους ώστε να βελτιώσουμε την διακυβέρνηση στο Αφγανιστάν. Θα έχουμε και εκλογέ άλλωστε φέτο. Επομένω, στόχο μα θα πρέπει να είναι το να δημιουργήσουμε προποθέσει ε, χρηστή διακυβέρνηση. Επίση, για τις σχέσεις ε, ΝΑΤΟ-ΕΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι εάν κάτσουμε να περιμένουμε τη λύση του Κυπριακού, περιμένουμε πάρα πολύ καιρό. Να βρούμε πρακτικές λύσεις πρακτικά μέσα πολιτικής. Και επίσης να λάβετε υπόψη τις σχέσεις Τουρκίας και πολιτικής ε, άμυνας και ασφάλειας. Διότι η Τουρκία θέλει να συμβάλλει περισσότερο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, όμως πάντοτε υπάρχουν φράγμοι, δεν σας δεν μπαίνω τώρα στις τα ξέρετε. Όλα αυτά παρακαλώ λάβετε τα υπόψη. Thank you, Mr. Vaid. I would like to hear something also about Cyprus, but you didn't say anything about that. So the floor is to Mr. Fugler from European Parliament. Ja, vielen Dank. Ich habe eigentlich nur eine sehr konkrete Frage. Ο κ. Φλούγκερ, ερώτηση. Όλο και περισσότερο στο στρατιωτικό επίπεδο ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ερώτηση λοιπόν, πώς το εκτιμάτε αυτό και σε ποιους συγκεκριμένους τομείς, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να γίνει αυτή η επέκταση και ποια συγκεκριμένη μορφή θα πρέπει να πάρει. Εγώ θεωρώ ότι αφενός έχει νόημα να συζητούμε για το μεγάλο στρατηγικό επίπεδο, από την άλλη μεριά είναι και σημαντικό να ανταλλάξουμε απόψεις και να ανταλλάσσονται και πληροφορίες <clears throat> στο στατιωτικό επίπεδο. Ποια είναι η θέση σας. Ε, well, thank ε, Ευχαριστούμε πολύ Λεωπρόεδρος. Και εγώ έχω μια ερώτηση σε σχέση με το πώς βλέπει η Ευρώπη τα πράγματα μια που τώρα η σημερινή συγκυρία προσφέρει κάποιες ε, ευκαιρίες. Έχουμε αυτές τις μεταβολές όπως την αλλαγή την κυβερνητική στις είπα οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω εσείς πώς τα βλέπετε πώς τα βλέπετε ως αυτό το θετικό σκέλος μπορούμε να έχουμε την ένταξη νέων χώρων προς τις Γαλλίες. Τι ρόλο επίσης μπορεί να παίξει η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας ή η καθυστέρησή της. Και έτσι αυτό να είναι ακόμα μια μεταβλητή στην ε, ασφαλειά μας Το ΝΑΤΟ είναι μια οργάνωση, από την άλλη μεριά εμείς δεν έχουμε οργάνωση, εμείς έχουμε μια πολιτική ασφαλείας. Άρα εσείς πώς τα βλέπετε, τι, τι, πώς μπορούμε να έχουμε κάποια εξέλιξη από πλευρά της Ευρώπης. Επίσης, άλλη μια ερώτηση όσον αφορά την οικονομική κατάσταση. Τι ευκαιρία μπορεί από εκεί να αναδεθεί. Πώς μπορούμε, επομένως και από αυτής της πλευράς, να βελτιώσουμε την κατάσταση από πλευράς ασφάλειας. Σας ευχαριστώ. Και έχετε το λόγο, γιατί δεν έχει ζητήσει άλλο το λόγο για ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις στη σειρά και όσο πιο γρήγορα μπορώ. για το θέμα των κοινοβουλευτικών επαφών και των επαφών με το Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το Ινστιτούτο σας έχει ήδη προχωρήσει σε κάποιες προτάσεις, έχει δημιουργήσει ένα κόκκους, όπως λένε μια ομάδα στήριξης στο εσωτερικό του Αμερικανικού Κογκρέσου, που εργάζεται εδώ και αρκετό καιρό και είναι ένα θετικό βήμα. θα μπορούσαμε ίσως να προσκαλέσουμε αυτές τις ομάδες στήριξης ή κάποια άλλα μέλη του Κογκρέσου, εν περιπτώσει, στις συναντήσεις κορυφής και πράγματι το Κογκρέσο θα πρέπει να συνδεθεί με τις προσπάθειές μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ίσως προσέξει στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάντα πολύ καλές σχέσεις βέβαια, αλλά η γραμματεία του Συμβουλίου δεν έχει κάνει τόσο καλή δουλειά στον τομέα αυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει ο Νταν κάτι σε αυτό αργότερα. Αλλά έπρεπε να το υπογραμμίσω. Για το Αφγανιστάν. Είναι αλήθεια, πρόεδρε, ότι έχουμε πολλές φορές διαφορετικές αντιλήψεις για τους κινδύνους και τους στόχους της αποστολής αυτής, με την εξαίρεση ένα-δύο κρατών στην Ευρώπη, έχουμε πάει εκεί σαν ένδειξη αλληλεγγύης ε, προς τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η αντίληψη ότι η ασφάλειά μας απειλείται από την κατάσταση στο Αφγανιστάν δεν υπάρχει. και δεν πρόκειται μάλλον και να αλλάξει σύντομα προς τη μία κατεύθυνση ή την άλλη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη προφανώς ανάλογα με την πολιτική άποψη που έχει ο καθένας. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να βελτιώσουμε την παρουσία μας εκεί. η αστυνομική δύναμη δεν πέτυχε. Απέτυχε πλήρως. Δεν έχει χρήματα, δεν έχει προσωπικό, είναι κλειδωμένη σε ορισμένα στρατόπεδα, δεν κάνει δουλειά. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα εδώ. Οι περισσότεροι Αυγανοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει. Πρέπει να γίνουμε πιο σοβαροί σε σχέση με αυτό και εγώ προσωρινά πιστεύω ότι η Γραμματεία του Συμβουλίου θα πρέπει να δει το θέμα του Αφγανιστάν με μεγαλύτερη σοβαρότητα γιατί δεν το έχει κάνει αυτό όσο θα μπορούσε. Αυτό που ακούω πάρα πολύ συχνά στη Washington είναι ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό αντιπρόσωπο για το Αφγανιστάν. Έχουμε ένα ειδικό ε, ε, εκπρόσωπο για το Αφγανιστάν που θα καλύψει όπου να είναι και το Πακιστάν Θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο του και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γόητρο έχει. Θέλουμε ένα Χόλμπροκ στο Αφγανιστάν. Κάποιοι στη Ουάσιγκτον μου έλεγαν ότι χρειαζόμαστε τον Πάτι Ashdown στο Αφγανιστάν. Τώρα για τα πυρηνικά και τη ρωσική πολιτική. Νομίζω ότι ακούστηκαν κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις. Το θέμα είναι σοβαρό, ιδιαίτερα από τη δική μας πλευρά, από πλευράς Ευρώπης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πιστέψουμε πράγματι ότι οι μειώσει στρατευμάτων από αμερικανικής πλευράς ε, θα αντιστοιχούν σε ανάλογες τέτοιες και από πλευράς των Ρώσων. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν έχουμε την εμπιστοσύνη ότι μια τέτοια διαδικασία θα πετύχει, είναι μια διαδικασία που πρέπει να την επιδιώξουμε και νομίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή χωρίς απαραίτητα να προηγηθούν σε βάθος διαβουλεύσεις. Για τον κύριο Λαντσμπέργκης, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας και για τα θέματα ορολογίας θα πρέπει να έρθω σε επαφή με τους συναδέλφους που έγραψαν το συγκεκριμένο κεφάλαιο εγώ δεν θα ήθελα εδώ να πω κάτι το μη σωστό. Υπάρχει διαφορά πάντως ανάμεσα στο CIS και στο NIS. Η Γεωργία δεν είναι μέλος του CIS, της Ομοσπονδίας, της Συνομοσπονδίας μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως εδώ να κάνω και λάθη, δεν τα ξέρω καλά. Για το αν θεωρούμε τώρα τη Ρωσία ότι ακολουθεί το δρόμο της δημοκρατίας. Προφανώς και το θεωρούμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η Ρωσία κινείται μακράν της δημοκρατίας προς ε, κάποια αυταρχικά ε, συστήματα ε, κρατικής διοίκησης και αυτό είναι αποσταθεροποιητικό στην περιοχή, είναι λυπηρό και ίσως το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα πρέπει να το λέει πιο ξεκάθαρα. Πάντως Αν αυτό σημαίνει τώρα ότι η ασφάλεια στην περιοχή μπορεί να καταστεί εφικτή χωρίς τη Ρωσία, η απάντησή μου εδώ δεν είναι τόσο σίγουρη. Η Ρωσία σίγουρα δεν είναι δημοκρατική. Σε αυτή τη φάση είναι πάντα εταίρος με τον οποίο πρέπει να συζητάμε, να κάνουμε πρακτικές συμφωνίες, για να βελτιώσουμε την ασφάλειά μας στην περιοχή. Γιατί η χρηστή διακυβέρνηση στο Αφγανιστάν. Πράγματι εκεί υπάρχει πολλή διαφθορά, η πολιτική του Καρζάη έχει απογοητεύσει πάρα πολλούς. Εμείς σε συνεργασία με τους εταίρους μας δεν ξέρω τι μπορούμε ακριβώς να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και να μην εμπλακούμε σε εσωτερικές διαφορές και διαφωνίες στο εσωτερικό του Αφγανιστάν. Πρέπει να βοηθήσουμε τη δικαστική εξουσία, τους δικαστές. Πάρα πολλοί από τους δικαστές της χώρας αυτής είναι αναλφάβητοι αλλά δεν μπορούμε να εμπλακούμε νομίζω στην αυγανική εσωτερική πολιτική. Για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και Τουρκία υποστηρίζω αυτά τα οποία είπατε. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό. Για τη γαλλική επιστροφή νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό σας συμβάν και σε επίπεδο πρακτικό και σε επίπεδο συμβολικό. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει κανείς τις σχέσεις της διατλαντικές, είτε είναι Ευρωπαίος, είτε είναι Αμερικανός, είτε είναι... έχει αλλάξει πολύ και με την επιστροφή των Γάλλων στο ΝΑΤΟ νομίζω ότι η συμβολική σημασία είναι πολύ μεγάλη αυτή της κίνησης. Η Γαλλία παραδοσιακά συμμετείχε βέβαια είναι μία από τις χώρες η οποία συμμετέχει περισσότερο στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ παρά ότι ήταν μακράν κάποιων μορφών συντονισμού και ε, λήψης απόφασης στο ΝΑΤΟ. Για την διοικητική δομή του ΝΑΤΟ, λοιπόν και σε συμβολικό και σε πρακτικό επίπεδο αυτό το οποίο έγινε ήταν ιδιαίτερα θετικό. Συγγνώμη υπάρχουν ίσως και θέματα στα οποία δεν μπόρεσα να δώσω απαντήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ζαμπορόφσκι, περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασής μας. για τις πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και τα πυρηνικά όπλα από τον Ιαν Άντωνη. Ο κύριος Άντωνη είναι υπεύθυνο συντονιστή τη ομάδα για την ε, μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και των όπλων μαζική καταστροφή στο ΣΥΠΡΙ στη Στοκχόλμη. Έχει κάνει πάρα πολλέ ε, μονογραφίε και έχει συγγράψει πολλά για τον έλεγχο των εξοπλισμών, το εμπόριο των όπλων και είναι συντονιστής της ομάδας για την αναθεώρηση της πυρηνικής πολιτικής του ΝΑΤΟ. Μια εξαιρετική μελέτη την οποία πήραμε και στη σοσιαλιστική ομάδα εκτιμούμε ιδιαίτερα τα έγγραφα του Σύπρη και τα χρησιμοποιούμε στις συζητήσεις μας τις οποίες κάναμε για τα πυρηνικά τον προηγούμενο Δεκέμβρη. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, όπως μας είπε και ο κύριος Χάμιλτον, μετά από τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου Ομπάμα και του Προέδρου Σαρκοζή. Κύριε Άντωνη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, όχι πάνω από 10 λεπτά, για να γίνει συζήτηση. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να είμαι ανάμεσά σας σήμερα. Είναι τιμή για μένα που, σας, ε, που είμαι μαζί σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και στις προκλήσεις τις οποίες παρουσίασε ο Ντάν σχετικά με το θέμα των ε, πυρηνικών δυνάμεων μικρής εμβέλειας στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε εδώ και αρκετά ε, χρόνια, αρκετούς μήνες μάλλον, σε συνεργασία και με Ινστιτούτα Γερμανικά Κανονικά ε, εφόσον έχουν λειτουργήσει τα πρακτικά θα πρέπει να έχετε κάποιο σημείωμα από πλευράς μου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται με τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων γενικότερα. το πλαίσιο της συζήτησης για τις πυρηνικές δυνάμεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ έχουμε δυνάμεις των ΗΠΑ, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουν τα τελευταία 10 με 15 χρόνια περάσει από πολλές διαδικασίες εξορθολογισμού με βάση τις συζητήσεις που είχαμε και με την Διεθνή Γραμματεία του ΝΑΤΟ και με τις, τα Υπουργεία. Από ό,τι φαίνεται το ΝΑΤΟ βραχυπρόθεσμα δεν θα σταματήσει να είναι μια πυρηνική συμμαχία. Σχετικά με τα συστήματα μικρής εμβέλειας υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό αυτών των όπλων, μικρού βεληνικούς, τα οποία είναι αποθηκευμένα στην Ευρώπη, σε διάφορες χώρες. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν τέτοια όπλα στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Τουρκία. Ίσως και να υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, από ό,τι φαίνεται όμως έχουν απομακρυνθεί και δεν πρόκειται να επιβεβαιωθεί τίποτα γύρω από αυτό. Ίσως επίσης η Ελλάδα να συμμετέχει σε κάποιες τέτοιες πυρηνικές ε, από κοινού προσπάθειες αν και δεν είναι σαφές κάτι τέτοιο. Σχετικά με τα συστήματα λοιπόν μικρού βεληνικούς, το ΝΑΤΟ έχει αναλάβει την υποχρέωση να διατηρεί επαρκείς δυνάμεις στην Ευρώπη. Αυτή η υποχρέωση όμως είναι εξαρτημένη από το αν οι δυνάμεις αυτές ανταποκρίνονται σε ορισμένα κριτήρια. Ευελιξία, επιβιωσιμότητα, έτσι ώστε οι δυνάμεις αυτές να είναι αξιόπιστες και αποτελεσματικές στα πλαίσια της προσπάθειας αποτροφής πολεμικών συγκρούσεων. Με τα χρόνια και με την εξέλιξη της τεχνολογίας αυτά τα χαρακτηριστικά επιβιωσιμότητας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας έχουν τεθεί σε αμφισβήτηση. Έχουμε προχωρήσει σε μια αναθεώρηση της πολιτικής του ΝΑΤΟ και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Η συζήτηση γίνεται παράλληλα και στη ΗΠΑ, όπως υπόθηκε, και ίσως να οδηγήσει σε κάποια πρώτα αποτελέσματα στις αρχές του 2009, στα τέλη του 2009, αρχές του 2010. Η συγκυρία η χρονική λοιπόν είναι πολλά, προσφέρει πολλά σε αυτή τη φάση. Κάποιες άλλες πλευρές της πολιτικής της νατοικής, τις οποίες θα πρέπει να δούμε, και πέρα από τα θέματα της αξιοπιστίας και της ελαστικότητας, της ευελιξίας μάλλον, η άποψη του ΝΑΤΟ βασίζεται στην ισότητα της κατανομής των βαρών και στην αρχή της αλληλεγγύης. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου τα πυρηνικά όπλα ήταν πολύ μεγαλύτερα σε αριθμούς εννοώ και είχαν κατανεμηθεί σε πολύ περισσότερες ε, σύμμαχες χώρες. Οι πυρηνικές δυνάμεις έχουν θα έλεγα αναδιπλωθεί από το 1991 από τότε έχουν υπάρξει βασικές αλλαγές και σε αριθμούς και στους τρόπους ανάπτυξης. Λιγότερες χώρες συμμετέχουν και αντί να υπάρχουν 13 ή 14 μορφές όπλων τώρα έχουμε μία μορφή. Αυτά τα θέματα λοιπόν αλληλεγγύης και κατανομής του βάρους είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Έχουν γίνει αναφορές και στο γενικότερο περιβάλλον για τον έλεγχο των όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχω καλυφθεί εδώ από τους προηγούμενους. Αυτό πάντως είναι ένα θέμα το οποίο ε, δείχνει ότι για το ΝΑΤΟ ισχύουν οι ειδικέ συμβάσεις και οι ειδικέ υποχρεώσεις σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο των Εξοπλισμών. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η εντολή για τη διαπραγμάτευση με τη Ρωσία όταν ξεκινήσει εκ νέου η συζήτηση για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, αλλά από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη φάση υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας για τις πυρηνικές δυνάμεις που είναι εκτός διεθνών συμφωνιών. Από το ΝΑΤΟ έχουμε 500 όπλα, 400 στην Ευρώπη και 100 ε, μπορούν μέσω πυράβλων κρούζ ή υποβρυχίων να ε, εκτοξευθούν από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και έχουμε 2.000 αντίστοιχα όπλα τουλάχιστον από πλευράς ρωσικής. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς εφαρμόζουν τις πολιτικές ανηλυμένες υποχρεώσεις τις οποίες εξέφρασαν το, ε, από το 1991 και μετά Πάντως αυτά τα πυρηνικά όπλα μικρού βεληνικούς είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Στο λίγο χρόνο τώρα που έχω θέλω να θέσω κάποια επιπλέον θέματα αλλά με πολύ τηλεγραφικό τρόπο, συνοπτικό τρόπο χωρίς λεπτομέρειες. Το βασικό που θέλω να πω είναι ότι τα, τους επόμενους 10 με 12 μήνες υπάρχει λόγος για να δούμε αν πραγματικά θα πρέπει να παραμείνει η πυρηνική αποστολή του ΝΑΤΟ υπό τη μορφή που έχει σήμερα ή αν θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και ποιες θα είναι αυτές. Ξέρετε ότι έχουμε ξεκινήσει για την παραγωγή ενός εγγράφου που αφορά τη νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ και υπάρχει ένα κεφάλαιο για την πυρηνική πολιτική του ΝΑΤΟ. Ε, φυσικά θα μπορούσαμε να μην προτείνουμε κάποιες αλλαγές και να χρησιμοποιήσουμε και την ίδια ορολογία. Το ΝΑΤΟ δηλαδή να κάνει μια δήλωση απλά ότι τα πυρηνικά όπλα είναι απαραίτητα σήμερα, στο άμεσο μέλλον και γενικότερα στο αόριστο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε γιατί χρειαζόμαστε τα πυρηνικά όπλα και τι ρόλο παίζουν τα πυρηνικά όπλα. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό στα πλαίσια της αξιολόγησης των απειλών και εδώ υπάρχουν ορισμένα μηνύματα τα οποία είναι σχετικά θα έλεγα αρνητικά στην περιφέρεια της διαβρωμένης συμμαχίας, διευρυμένης συμμαχίας. Υπάρχουν χώρες που αποκτούν νέες τεχνικές δυνατότητες στρατιωτικές και σε επίπεδο ε, πυράβλων και σε επίπεδο μέσων χρήσης των πυράβλων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές στη συμπεριφορά των χωρών οι οποίες ε, χρησιμοποιούν ε, τα πυρηνικά όπλα και τα όπλα γενικότερα. Το περιβάλλον απειλών δηλαδή είναι ένα περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ε, αυτό αφορά χώρες όπως και η Συρία. Το θέμα είναι πώς οι δυνάμεις αυτές οι πυρηνικές μικρού βεληνικούς θα μπορέσουν να καταπολεμήσουν τις υπάρχουσες απειλές τα παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιήσαμε ε, είδαμε ότι οι πυρηνικές αυτές δυνάμεις δεν βοηθούν ιδιαίτερα. Και έχουμε κάποιες εμπειρίες από τον πρώτο πόλεμο στον Περσικό κόλπο σαν παράδειγμα όπου είχαμε κάποιες ενδείξεις από τη δεκαετία του 80 για κάποια όπλα μαζικής καταστροφής Έγιναν αναφορές επίσης και για το τι συμβαίνει στα σύνορα ανάμεσα στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν όπου ήδη υπάρχει μια χώρα πυρηνική δύναμη η οποία διεξάγει επιχειρήσεις στο εσωτερικό μιας άλλης πυρηνικής χώρας όπως το Πακιστάν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της συγκεκριμένης χώρας. Προς το παρόν τα πυρηνικά όπλα δεν έχουν παίξει κάποιο θετικό ή αρνητικό ρόλο στην εξέλιξη της κρίσης. Το ίδιο ισχύει και σχετικά με το Ιράν. Ε, προφανώς η ύπαρξη δυναπίθανος κάποιων πυρηνικών δυνάμεων ε, μεγάλου βεληνεκούς είναι κάτι το θεωρητικό. Και δεν ξέρουμε ακριβώς ε, αν θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορούν να παίξουν οι δυνάμεις αυτές μικρού βεληνεκούς κάποιο ρόλο στην περιοχή. Υπάρχουν και τεχνικά θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σχετικά με τα συστήματα εκτόξευσης τα οποία χρησιμοποιούνται ανάμεσα στις χώρες οι οποίες συνεργάζονται. Πριν, από, κατά τη διάρκεια του πολέμου υπήρχαν πάρα πολλά συστήματα, ενώ τώρα έχουμε μόνο ένα σύστημα, την εκτόξευση από αεροσκάφη. Ο στόλος ο οποίος χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα θα μπορεί να πετά ως έχει μέχρι το 2020-2025 αλλά για την Ευρώπη γύρω στο 2012 με 2015 θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τον εξυγχρονισμό των συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, δηλαδή τα IDV, Tornado κτλ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύστημα διάδοχο το οποίο να έχει επιστοποιηθεί. Το F-35, το JDF-SF δεν έχει επιστοποιηθεί για πυρηνικές αποστολές το F-22 Raptor ούτε και αυτό έχει πιστοποιηθεί για μεταφορά πυρηνικών όπλων, οπότε οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες για να κάνουν τροποποιήσεις και να προτείνουν νέα συστήματα εκτόξευσης. Ίσως θα πρέπει να βρούμε και εναλλακτικέ λύσεις, πυράβλους από το έδαφος που να εκτοξεύονται από το έδαφος. Θα πρέπει να υπάρξουν πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Υπάρχει το γαλλικό σύστημα επίγειας εκτόξευσης που είναι κομμάτι του γαλλικού συστήματος αποτροπής αλλά η Γαλλία διευκρίνησε ότι αυτή τη στιγμή μπουν στο ΝΑΤΟ τα πυρηνικά θα μείνουν εκτός πλήρους συμμετοχής. Όλα θα τα συζητήσουν εκτός από τα πυρηνικά όπλα. Έχουμε λοιπόν πρακτικά ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να, στα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αν δει κανεί λίγο και τις πολιτικές διαστάσεις, αναφέρθηκα ήδη στην κατανομή του άχθους, του βάρους, όχι μόνο λιγότερες χώρες συμμετέχουν στις πυρηνικές αυτές επιχειρήσεις σε σχέση με τον αριθμό των χωρών της διαβεμένης συμμαχίας, αλλά υπάρχουν και όρια στον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν. Τα όπλα όπως είπα αποθηκεύονται σε συγκεκριμένους χώρους αλλά δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλους χώρους. Στις νέες χώρες που είναι πιο κοντά στη Ρωσία γιατί έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να μην το κάνουμε αυτό στα πλαίσια της πρώτης συμφωνίας ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ρωσία. Υπάρχουν επίσης δυνητικά δυσκολίες και για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα όπλα από το ΝΑΤΟ σε κάποια σενάρια τα οποία δύσκολο μπορεί κανείς να μην φανταστεί. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου είχαμε κάποια ολοκληρωμένα στρατηγικά στρατιωτικά προγράμματα και η εφαρμογή του στην ουσία ήταν κάτι το οποίο αναλάβαναν σαφέστατα οι στρατιωτικές δυνάμεις, η στρατιωτική πλευρά. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο προγραμματισμός ε, εδώ γίνεται αντικείμενο συζήτηση σε όλες τις φάσεις. Υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης των συστημάτων και της χρήσης των συστημάτων και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των ιδίων. Αυτό θέτει πολλούς περιορισμούς στη χρήση των πυρηνικών όπλων σε οποιοδήποτε σενάριο ακόμα και στις πιο εκτεθειμένες χώρες της Συμμαχίας. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Τουρκίας που θεωρείται εκτεθειμένη. Είναι δύσκολο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις στρατιωτικές βάσεις της Τουρκίας για παραδοσιακές επιχειρήσεις, παραδοσιακές συμβατικές εννοώ, όχι πυρηνικά όπλα. Καταλαβαίνετε ότι αν το ζητούσαμε αυτό για αποστολές με πυρηνικά όπλα, το πρόβλημα θα ήταν πολύ σοβαρότερο. Ένα άλλο θέμα είναι ότι αν δεν είχαμε τα όπλα τι θα συνέβαινε. Νομίζω ότι κάποιες από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις έχουν συζητηθεί στο παρελθόν, δηλαδή διαφορετική παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο προχωρά το ΝΑΤΟ σε κοινέ ασκήσεις, περαιτέρω ειδικότερε εγγυήσει στις περισσότερο εκτεθειμένες χώρες και αναφέρομαι εδώ στις διμερείς συμφωνίες Ηνωμένων Πολωνίας, για την βελτίωση της συμμετοχής των χωρών αυτών στα πλαίσια της πυραυλικής άμυνας. Ανάπτυξη των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και αυτό είναι ένα κομμάτι του πακέτου των θεμάτων τα οποία ε, μπορούν να βοηθήσουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ και πέραν της ε, χρήσης πυρηνικών όπλων. Εν πάση περιπτώσει, τα λέω πολύ συνοπτικά και γρήγορα. Είναι σαφής η διαστάσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στο μέλλον στον τομέα των πυρηνικών όπλων. Υπάρχουν όμως και κάποια επιμέρους προβλήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει τους επόμενους 12 μήνες γιατί το 2010 θα υπάρξει αναθεώρηση μέσω της παγκόσμιας διάσκεψης της συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το τι θα ακολουθήσει το 2010. Αυτό το οποίο υποστηρίζω είναι ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να προχωρήσει στις συζητήσεις αυτές χωρίς προκαταλήψεις, να δούμε τι έγινε τα τελευταία 50 χρόνια, να δούμε ότι τα τελευταία 15 μάλλον χρόνια έχει τροποποιήσει τις πυρηνικές του ικανότητες με πολύ ε, σημαντικό τρόπο και ότι δεν έχουμε καμία ιδεολογική θα έλεγα αγάπη ε, προς τα πυρηνικά όπλα σαν ΝΑΤΟ. Πρέπει να είμαστε δεκτικοί, να πούμε ότι θα κρατήσουμε τα όπλα αν μας χρειάζονται, αλλά να πούμε επίσης ότι αν δεν μας χρειάζονται θα πρέπει να τα απομακρύνουμε. Ευχαριστώ, πάρα πολύ, δόκτωρα. Έχετε τώρα το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Ο κ. Ζαμάλφα από την Ιταλία. Ευχαριστώ. Μήπως θα μπορούσε ο κύριο ε, Άντωνη να συμπληρώσει τα όσα ενδιαφέροντα μα είπε στην εισήγησή του με το να μα ε, δώσει μια ε, εικόνα του τι γίνεται στην Ρωσία προ στρατηγικής για τα πυρηνικά. Οποιαδήποτε όπλα πυρηνικά μεσαίου, μικρού, μεγάλου βεληνικού. Πρόεδρο, χωρί μικρόφωνο. ναι. Ε, αυτά τα πυρηνικά, τα τακτικά πυρηνικά όπλα είναι ένα ζήτημα σημαντικό το οποίο συχνά ανακύπτει. Και σας ε, υπενθυμίζω ότι υπάρχουν κάποια α, δημοσιεύματα για τα πυρηνικά τα οποία έχουν αναπτύξει στην περιοχή του Καλίνιγκραντ. Οπότε και εγώ τώρα έρχομαι στο επόμενο θέμα. Μήπως θα ήταν δυνατόν να μπορέσουμε να έχουμε μια ρύθμιση για αυτά τα πυρηνικά όπλα, ούτως ώστε να καλύπτονται ε, ακριβώς όπως έγινε και με την ε, συνθήκη για τα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 τι γίνεται με αυτά τα ποινικά που ήταν να αποσυρθούν ε, υπάρχουν τελικά χρησιμοποιούνται ή όχι γιατί αυτό αποτελεί κίνητρο ή αντικίνητρο χρήσης ανάλογα The floor is to Mr. from Turkey. Ο κύριος Ερδέν από την Τουρκία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να κάνω ένα σχόλιο για τις βάσεις στην Τουρκία. Οι βάσεις στην Τουρκία χρησιμοποιούνται ευρέω για διάφορες επιχείρησει. Θα θυμάστε ότι στον πρώτο πόλεμο του Περσικού η, κυρίως η ε, βάση του Ιντσιρλίκ χρησιμοποιήθηκε από τους Αμερικανούς και για λογιστικές, δηλαδή για επιμελητία κλπ. αλλά και για να προστατευτεί το Βόρειο Ιράκ κατά του Σαντάμ. και ούτω ή άλλω και πάλι χρησιμοποιήθηκε η βάση του Ινσυρλίκα από τι δυνάμει τότε για να προστατεύσουν το βόρειο Ιράκ, του Κούρδου. Τώρα, η περισσότερη επιμελητία περνάει από την Τουρκία πάλι για τι δυνάμει του Ιράκ και για το Αφγανιστάν. Από τι βάσει τη Τουρκία περνάνε. Χρησιμοποιείται λοιπόν Εβραίο στην περιοχή. Σχόλιο λοιπόν αυτό. Τώρα, δεύτερο, όταν μιλούμε για πυρηνικά όπλα, έρχεται στο μυαλό μας το Ιράν. Για όλους είναι μεγάλη ανησυχία και ιδία για την Τουρκία. Βεβαίω η Τουρκία είναι απολύτως αντίθετη στην ιδέα το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό εξοπλισμό, πυρηνική ικανότητα. Γιατί τότε βέβαια ε, θα ανατραπεί ο συσχετισμός δυνάμεων στην περιοχή. Έχω μια ερώτηση που ίσως είναι και άσχετη, δεν ξέρω. Είναι δυνατόν να γίνει μια πιο σε βάθος προσέγγιση, να ζητηθεί από το Ισραήλ να καταργήσει την πυρηνική ικανότητα που έχει και ταυτόχρονα να ζητηθεί από το Ιράν να μην αποκτήσει η πυρηνική ικανότητα και να αναγνωρίσει το Ισραήλ και το Ιράν και άλλες χώρες. Ίσως να είναι αφελής η ερώτηση αλλά αυτό σκέφτομαι. Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της περιοχής δηλαδή με ένα ενίο τρόπο, αντί να ασκείται μόνο στο Ιράν. Γιατί το Ιράν λέει, η Ινδία, το Πακιστάν και το Ισραήλ έχουν πυρηνική ικανότητα. Γιατί τη στερείται από εμά. Εγώ έχω μιλήσει πολύ με Ιρανούς και αυτό είναι το επιχείρημά τους. Ε, τι νομίζετε λοιπόν σχετικά με την προσέγγιση που ανέφερα. Κύριε Μπουβάρ. Ε, ε, σας ευχαριστώ. Δόκτωρ Άντωνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, εισήγησή σας και θα ήθελα ένα πράγμα μόνο να αναφέρω. Μας αν είπατε ότι η Γαλλία κάνοντας μια ιστορική αναδρομή ότι έχει την απόλυτη κυριαρχία όσον αφορά τα πυρηνικά. Δεν νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι Αμερικανικοί, Αμερικανοί εταίροι μας θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο περιορίζει τον προστατελισμό της Γαλλίας γιατί ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τη ΣΥΠΑ οι ένοπλες δυνάμεις αμερικανικές έχουν εθνικό χαρακτήρα και ουδέποτε, ουδέποτε ε, υπό ηγεσία νατοική και όταν ε, ζήτησε ο στρατηγό να λοιπόν, πούνε πόσε ποινικέ σκευές βρίσκονται σε γαλλικό έδαφο, πριν δηλαδή αποχωρήσει από το στρατηγικό σκέλο η Γαλλία. Ο Αμερικανό στρατηγό απέντησε στο στρατηγό Ντεγκόλ, λυπάμαι πολύ στρατηγέ, δεν μπορώ να σα το πω, είναι μυστικό. Και ο στρατηγό Ντεγκόλ του είπε, παρακαλώ, πρέπει να μάθετε ότι είναι η τελευταία φορά που ένα Αμερικανό στρατηγό λέει στον αρχηγό του Γαλλικού κράτου ότι μπορεί να απαντήσει από αυτού. Και για αυτόν τον λόγο ε, αποφάσισε ο στρατηγό να βγάλει από το στρατηγικό σκέλος του ΝΑΤΟ την ε, Γαλλία. επομένω, δεν θα πρέπει τώρα να υπάρχει μια σύγχυση ότι δηλαδή ε, το ότι ελέγχουμε πλήρω τις πυρηνικέ μας κεφαλέ δεν σημαίνει ότι δεν υπαγόμεθα στο επιτελείο, στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ. Ο κ. Φλούγερ είναι πολύ έβυχα αυτά τα δραματουργικά όταν αναφέρεστε σε, στο γαλλικό πυρηνικό οπλοστάσιο διότι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση οι Γάλλοι με το πυρηνικό του οπλοστάσιο η δική μου θέση είναι ότι τα πυρηνικά όπλα οφείλουν να καταργηθούν. Το ίδιο λέει και η συνθήκη της μη διασποράς. Και στις συζητήσεις εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε ασκούνται όλοι σε αυτοσυγκράτηση όταν τέθεται θέμα ε, πυρηνικών όπλων Γάλλων ή Βρετανών. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει για το Ιράν. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι σωστό να δακτυλοδεικτούνται πάντοτε οι άλλοι. Σωστό είναι να καταργηθούν όλα τα πυρηνικά όπλα. Και γι' αυτό η ερώτησή μου προς εσάς, κύριε Εμπειρογνώμων, τι λέτε για τον ρόλο του γαλλικού και βρετανικού πυρηνικού οπλοστασίου μέσα στα πλαίσια της ε, σχέσης με την άλλη ακτή του Ατλαντικού. Στη Γερμανία έχουμε ένα ιδιαίτερο συσχετισμό. Υπάρχει μια πυρηνική συμμετοχή. Δηλαδή η Γερμανία η ίδια δεν διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο αλλά έχει εντό εισαγωγικών συμμετοχή σαν να έχει μερίδιο στο αμερικανικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Εγώ βρίσκω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού. Εγώ πάντως είμαι απολύτως υπέρ κατεπηγόντως να εγκαταλείψει αυτή τη συμμετοχή η Γερμανία να αποχωρήσουν τα πυρηνικά όπλα των Αμερικανών από το γερμανικό έδαφος. Για μένα είναι ενδιαφέρον που βλέπω ότι στο έγγραφο των κυρίων Νάουμαν και Τσαχικασουίλη διατυπώνεται το πρώτο πλήγμα, το πρώτο πυρηνικό πλήγμα ως ενδεχόμενη επιλογή του ΝΑΤΟ. Ποια είναι η δική σας θέση. Αρχικά είπατε ότι υπάρχουν τόσα περίπου πυρηνικά όπλα, κεφαλές. Και αυτό είναι και ένα από τα κεντρικά προβλήματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, ούτε πού είναι σταθμευμένα τα όπλα αυτά, ούτε και πόσα είναι σε αριθμό. Έχετε κάποια ιδέα αν και πότε θα έχουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες γιατί αυτό είναι πολιτικά καυτό το θέμα. Και τέλος βρίσκω ότι είναι κεντρική σημασία στο θέμα εάν θέλει η ευρωπαϊκή πολιτική να είναι και αξιόπιστη να κάνει ίδια κάτι στο θέμα του πυρηνικού εξοπλισμού, στο θέμα του αφοπλισμού μάλλον και κυρίως βεβαίως και πρωτίστως στο θέμα του πυρηνικού αφοπλισμού. Γκόμες, αν δεν θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο, να τον λάβω εγώ. Και να υποστηρίξω την ερώτηση του Τούρκου συναδέλφου μας, διότι θεωρώ, φοβούμε, ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα σημείο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, όπου δεν θα μπορούμε να αγνοήσουμε το περιφερειακό αυτό πλαίσιο. Και είναι γεγονός ότι υπάρχουν πυρηνικές δυνάμεις στην περιοχή και εκτός της Ινδίας και του Πακιστάν και εννοώ το Ισραήλ νομίζω ότι το περιφερειακό πλαίσιο δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί και με την έννοια ότι βεβαίως το Ιράν κινείται προς την απόκτηση στρατιωτικής πυρηνικής ικανότητας και αυτό συμπαρασύρει και άλλες χώρες να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό μια αποπυρηνικοποιημένη ζώνη της Εγγύης Ανατολής θεωρώ ότι είναι απαραίτητη. Εάν δούμε κίνηση από πλευράς Αμερικανικής κυβέρνησης Ομπάμα, εγώ θυμούμαι στην τελευταία κοινοβουλευτική συνέλευση, νομίζω ήταν η πρώτη τελευταία συνάντηση στην ε, Ισλανδία, που αρχίσαμε να συζητούμε την αναθεώρηση της στρατηγικής αντίληψης και νομίζω η Νορβηγία έθεσε το θέμα ότι είναι ανάγκη δηλαδή να ξανασκεφτούμε το δόγμα του, της πυρηνικής αποτροπής Θυμάμαι ότι πολύ λίγοι τότε εξέφρασαν ανησυχίες ή επιφυλάξεις. Ελπίζω με τη νέα προσέγγιση της ε, κυβέρνησης Ομπάμα και μάλιστα και με αυτά τα σημαντικά άρθρα που ε, δημοσίευσαν Κίσιγκερ, Νάν, Σούλτς και Πέρι, ελπίζω ότι θα αντιληφθούν και περισσότεροι το άχρηστο των ε, πυρηνικών όπλων, για να πω ότι είναι το λιγότερο άχρηστα. Εγώ θέλω να πω και ε, θα ήθελα να ακούσω την άποψη του κ. Άντωνη ότι οι αντιστάσεις προέρχονται κυρίως από τις δύο πυρηνικέ ευρωπαϊκές δυνάμεις, Βρετανία και Γαλλία. Και εδώ υπάρχει και ένα τεράστιο έλλειμμα εδώ, με την έννοια ότι δεν τους αμφισβητούμε εμείς. Η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας δεν θέτει καν θέμα ότι υπάρχουν δύο χώρε με πυρηνικό οπλοστάσιο. Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν, Ιδιαίτερα τώρα, στο πλαίσιο αυτής της βαριάς οικονομικής κρίσης, όπου διαπιστώνονται τρομερά ελλείμματα και προσθέτεται αυτά και στα ελλείμματα των προϋπολογισμών άμυνας ή εξοπλισμών και χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές οι οποίες βεβαίω δεν αντιμετωπίζονται με πυρηνικά οπλοστάσια. Δεν θεωρείτε ότι θα είναι μια σημαντική ευκαιρία ώστε και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και όλοι μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αλλά και στα άλλα πλαίσια και στα πλαίσια της ε, ε, συνθήκης μη διασποράς να ξανασκεφτούμε τη στρατηγική και εν πάση περιπτώσει να αποφασίσουμε να καταργήσουμε τα πυρηνικά όπλα. Δόκτωρ. Σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Για να πάμε στην αρχική ερώτηση όσον αφορά το ρωσικό ποινικό προστάσιο. Έχει δίκιο ο Συνισκεύης ότι είναι πάρα πολύ βασικό θέμα. Δεν ε, ε, ανησυχώ για το κατά πόσον ε, έχουν τη θέληση Αμερικανοί να ασχοληθούν με αυτό με σχετικές συνομιλίες γιατί είναι κάποιοι που τους γνωρίζουμε, με έχουν ικανότητες είναι οι κατάλληλοι ε, άνθρωποι οι οποίοι συνομιλούν με την ρωσική πλευρά στην οποία τα πράγματα είναι τόσο σαφή. Ε, έχουν γίνει κάποιες ε, αλλαγές στην πολιτική του τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα προσθέσει περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση η Ρωσία όσον αφορά την ποινική αποτροπή σε σχέση με τον πρώτο προσθέσμα του προ τι συμβατικέ δυνάμει. Επίση, βλέπουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση στη Ρωσία πάρα πολύ σοβαρά βλέπει το να ε, κάνει μια μεταρρύθμιση στο, στο, στους ενόπλες Και κλείστηκε κάποια συμφωνία ε, ότι δηλαδή δεν θα θυγούν κάποια κεκτημένα του, του κα, κατεστημένου σε σχέση με το να μπορέσουν να να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια η πολιτική στα, του προσανατολισμού της στρατηγικής. Βέβαια είναι και θέμα έλλειψης διαφάνειας. Μπορούμε βέβαια να πούμε ότι έχουμε περίπου 10.000 πυρηνικά στον κόσμο, τα οποία έχουν αναπτυχθεί τώρα, είναι ενεργά. αν βάλουμε όλα αυτά τα οποία είναι και σε αποθήκες, πάμε στις 20.000. Είπα και η Ρωσία έχουν το 90% αυτών των πυρηνικών όπλων λίγο παραπάνω από τα μισά είναι τα ρωσικά. Όταν όμως κοιτάξει κανείς πιο συγκεκριμένα είναι δύσκολο κανείς να είναι βέβαιος για οτιδήποτε όσον αφορά ιδίω τα όπλα μικρού βελνικούς της Ρωσίας. Όπως ξέρετε τώρα το πόση διαφάνεια υπάρχει εξαρτάται από το πώς πάνε οι συνομιλίες οι με τα πυρηνικά στην Ευρώπη τον ΝΑΤΟ τα θέλουμε, τα καταργούμε. Θα μπορούσαν επίση να αρχίσουν συνομιλίε με του Ρώσου για να κατεβούν σε κάποια συμφωνία ενδεχομένω. Ε, Α πούμε να έχουμε κάποιο είδου πολιτικέ δεσμεύσει σε σχέση με τα νέα κράτη-μέλη και να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Και έτσι ε, σε αντάλλαγμα να έχουμε διαφάνεια από πλευρά Ρώσων. Και έτσι να είμαστε πιο βέβαιοι, να μπορούμε να ξέρουμε ποιες είναι οι παράμετροι του προβλήματος. Όσον αφορά τώρα το Ιράν, αλλά και το Ισραήλ, ο πλευράς της ε, Ιρανικής πολιτικής, οι μεταβλητές σημαντικές είναι οι διμερείς σχέσεις του Ιράν με τη ΣΥΠΑ. Όμως, από πλευρά Ιράν πάλι, είναι και θέμα περιφερειακής ασφάλειας. Η Ευρώπη φυσικά και δεν μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ, αλλά μπορεί να διευκολύνει, να διευκολύνει τις επαφές όσον αφορά την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία παίζει υποδηματικό ρόλο το οποίο επίσης συνδέεται και με την υπόθεση των πυρηνικών. Εάν θέλουμε στο μέλλον αυτά να ισχύσουν στα πλαίσια των σχέσεων μας με το Ιράν για την πυρηνική αποτροπή, τότε θα προσέξουμε να μην έχουμε μια σχέση ανταγωνισμού. Όμως ε, ιστορικά δεν υπάρχει έχθρα όπως υπάρχει έχθρα ιστορικά μεταξύ Ιράν και Τουρκίας, Ιράν και Ισραήλ. Άρα γιατί να προχωρήσουμε σε μια κίνηση που θα τους θέσει όλους αντιμέτωπους προς αλλήλους. Ιστορικά προκύπτει ότι υπήρχε ε, μεταξύ ε, Ιράν, Ισραηλινών ε, μια συμμαχία, είχαν κοινό εχθρό τους Άραβες. Άρα θα πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά οι Ευρωπαίοι τι ρόλο θα παίξουν. Τώρα το θέμα των ε, σχέσεων Γαλλίας και ΝΑΤΟ δεν διαφωνώ με τίποτα πώς άκουσα. Το θέμα είναι πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μία, ε, ένα προβληματισμό εάν δεν συμμετέχει η Γαλλία. Καλά, θα, πάντα υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις ad hoc, αλλά φυσικά είναι πιο εύκολο αν κανείς ε, συμμετέχει άσχετα από την υπαγωγή στο αρχηγείο, τουλάχιστον μπορεί να γίνουν συζητήσεις. Ο ρόλος τώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, των Γαλλικών Πυρηνικών σχέσεων με τις διατλαντικές σχέσεις, να το δούμε έτσι ευρύτερα, αυτό δεν αλλάζει το παγκόσμιο σκηνικό του, τι θα γίνει όσον αφορά την ανάπτυξη, τι θα γίνει με το μέλλον των πυρηνικών από πλευρά Γαλλία και Αγγλία, θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Σήμερα κάποιε χώρε όπω η Ινδία έχουν φτάσει σε κάποια πολύ προχωρημένα στάδια του να κατασκευάσουν ε, πυρηνικά υποβρύχες δοκιμές, εκτοξεύσεις ε, πυράβλων, προγράμματα. Έχουν προχωρήσει πολύ. Η δε Κίνα Επίσης εξυγχρονίζει τις ε, ενόπλες δυνάμεις. Και θεωρείται αυτό το, το ελάχιστο μπορεί να γίνει, το να έχουν δηλαδή ένα τέτοιο πλωστάσιο. Έτσι, έτσι δείτε τα πράγματα και όχι ε, καθαρά ε, διατλαντικά. Τώρα, το τελευταίο σημείο είναι ότι χρειάζεται να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά αυτά τα στρατηγικά όπλα σε επίπεδο διμερές, τι γίνεται μεταξύ ΙΠΑ και Ρωσίας. Χρειάζονται όλα αυτά, αλλά χρειάζονται όλα μαζί. Δεν υπάρχει βήμα, δεν υπάρχει πλατφόρμα για να συζητηθεί το θέμα αυτό από όλες τις χώρες που έχουν οι, μεγάλοι, οι πέντε μεγάλοι, η Ινδία και το Πακιστάν δηλαδή Ρωσία, Αμερική, Ινδία, Ιράν, Πακιστάν. Ε, και έτσι μπορούμε να δούμε την ευρύτερη εικόνα, ούτω ώστε να θεωρήσουμε ότι όλοι μπορούν στο ίδιο τραπέζι πέραν των διμερών επαφών. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθηγητά, λέει πρόεδρο. Οπότε τώρα ε, θα ήθελε ο συνάδελφος να δευτερολογήσει για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Άννα Μαρία. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σένα προσωπικά για τη σημερινή συνάντηση. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις και οι απόψεις που αντιλάγησαν. Ευχαριστώ τους ομιλητές λοιπόν. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ για την δραστήρια συμμετοχή τους και την αρκετά μεγάλη μάλιστα συμμετοχή τους στη συνάντηση αυτή. Θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε αυτά τα θέματα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες ο συνήθως ο πρόεδρος της ε, συνέλευσης αυτής θα απευθύνει το λόγο στη συνάντηση κορυφής στο Στρασβούργο και στο ΚΕΛ την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα μάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε κάποια από τα θέματα τα οποία συζητήσαμε σήμερα όπως οι δυνατότητες εξελίξεων της συμμαχίας μας σε αυτούς τους ε, δύσκολους χρόνους. Το βάρος της διατλαντικής μας συμμαχίας, όπως λένε και λέγω και εγώ, είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε σύμμαχοι και φυσικά στο ίδιο επίπεδο υπάρχει ανάγκη να εξετάσουμε εκ νέου τις νέες διαστάσεις της σχέσης μας και τη μεταρρύθμιση του ΝΑΤΟ. Να δούμε τη μεγάλη σημασία που έχει η παρουσία μας στο Αφγανιστάν. Θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι να γίνουν σοβαροί για το Αφγανιστάν και απαιτείται να υπάρξει και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. και να τονίσουμε και τον σημαντικό ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξουν οι κοινοβουλευτικοί στον τομέα αυτό γιατί εκπροσωπούν τους λαούς της Ευρώπης και με τη δική μας συνεισφορά μπορούμε να εξηγήσουμε καλύτερα τα προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά θα συνεισφέρουν στην διαδικασία μεταρρύθμισης της στρατηγικής αντίληψης του ΝΑΤΟ Βρισκόμαστε σε ένα πρόωρο στάδιο της επεξεργασίας των θέσεών μας αλλά νομίζω ότι οι συζητήσεις οι οποίες προηγήθηκαν ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει η κυρία Γκόμες, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Υποεπιτροπής Ασφαλείας, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που είναι μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ που ήρθαν εδώ σήμερα και που κατέστησαν τις συζητήσεις αυτές τόσο χρήσιμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες, τον Ταν Άμιλτον, τον κύριο Ζαμπορόφσκι και τον Ιαν Άντωνη. για πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, δηλώσεις και τα στοιχεία που μας έδωσαν. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να μάθουμε για να μπορέσουμε να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Όχι μόνο ότι είναι καθήκον μας αυτό, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι η σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ΝΑΤΟ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μέσω της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών ικανοτήτων θα συνεισφέρουμε και στην περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεων του ΝΑΤΟ και του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Ήταν ε, ουσιαστική συζήτηση που κάναμε ιδιαίτερα για τα πυρηνικά όπλα από τότε που είμαι εδώ εδώ και πέντε χρόνια είτε στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης είτε της Επιτροπής Ασφαλείας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον και νομίζω ότι οι τελευταίες εξελίξεις θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με μια στρατηγική αντίληψη πιο κατάλληλη. Υπάρχει και το θέμα της οικονομικής κρίσης. Η οικονομική κρίση επηρεάζει τις επιλογές μας στον τομέα της ασφάλειας και της κάλυψης των προβλημάτων. Έχουμε την ευθύνη εδώ να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις έτσι ώστε οι πολίτες μας να έχουν το καλύτερο value for money στη συγκεκριμένη περίπτωση της ασφάλειάς τους. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες.